What's the time? Good morning, dear colleagues. Καλή σας μέρα αγαπητοί συνάδελφοι, καλημέρες κυρίε και κύριοι. Είναι 9 ναι και 5, οπότε ας αρχίσουμε τη σημερινή μας συνεδρίαση. Είμαστε στα σημεία 8, 9, 10, 11 και 12. Είχατε χρόνο να τα πείτε, συνάδελφοι, τώρα δουλειά. Λοιπόν, είπαμε, περνάμε στα σημεία 8, 9, 10, 11 και 12, που είναι ψηφοφορίες. Και πρέπει να τις δεκτερώσουμε σε μία ώρα. Σημείο 8, λοιπόν. Θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτηση διεθνού προστασία που υποβάλλεται σε κράτο μέλο από επίκο τρίτης χώρα ή από απάρτιδα τα Πάτρινα. Πριν περάσουμε στην ψηφοφορία, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον εισηγητή, κυρία Μανέσκου. Ευχαριστώ. Θέλω πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέρφους από τις άλλες πολιτικές ομάδες για την τόσο καλή συνεργασία που είχαμε επί της γνωμοδότησης αυτής. Είναι η γνωμοδότησή μας προς τη ΛΥΜΠΕ που είναι η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή. Έχουμε διάφορες ε, τροπολογίες, οι περισσότερες έχουν να κάνουν βέβαια με τη Λίμπε. Θα δείτε που βάζω πλην, ακριβώς γιατί είναι θέμα της Λίμπε. Και από τις συζητήσεις που είχα με την εισηγήτρια της Λίμπε, μας είπε να ασχοληθούμε εμεί με ό,τι είναι δικιά μας αρμοδιότητα. Αυτό προσπάθησα λοιπόν να κάνω και στη, στον κατάλογο αυτό ψηφοφορίας. Δεν είναι ότι δεν είναι καλές οι τροπολογίες, αλλά αφού πρόκειται για θέματα λίμπε, δεν νομίζω ότι μας αφορούν. Τώρα κάποιοι συνάδελφοι ήδη έχουν υποβάλει τις τροπολογίες τους αυτές στην ίδια τη λίμπε, οπότε είναι εξασφαλισμένοι. Έχουμε και προφορικές τροπολογίες, που επίσης είναι αρμοδιότητα της ΛΥΜΠΕ, οπότε θα προτιμούσα να τις καταψηφίσουμε εμείς. Πρόεδρος, καλώς. Κύριε Χιμένες Μπαρότ. Δεν έχω την ε, κάρτα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Ήθελα να σας ενημερώσω γι' αυτό. Ε, στο Στρασβούργο φοβάμαι ότι έχει μείνει. Ωραία, τότε εσείς διανοτάσω στις χειρός. Καλώς, δεν ζητά κανένας άλλος το λόγο. Ωραία, τότε ψηφίζουμε. Από πού αρχίζουμε. Μάλιστα. Τροπολογία 52. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 53. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 54. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 55. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 56. Υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Πρέπει να μιλήσουμε και στο διευρυμένο πρόεδρο για αυτό. 57 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 58 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 59 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 60 υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται. 61-62 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 63 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 64 υπέρ. Να ελέγξουμε. Ωραία. Ελέγχουμε την 63 ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα τη φοφορίες απορρίφθηκε όντως. 64. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 65 μέχρι και 68 υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά, ψηφίστε. Πέρας της ψηφοφορίας, εγκρίθηκε. 69 υπέρ, όχι, εγκρίθηκε η προηγούμενη, οπότε καταπίπτει αυτή. Και φτάνουμε στις 74-75 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. 76 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. 77 υπέρ, α, αποσύρθηκε, μάλιστα. 78 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. 80 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 81 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 82 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 83-84 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. 85 με προφορική τροποποίηση. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 86 έχει αποσυρθεί. 87 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 88 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 89 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 90 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 91-92 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. 91-92 ψηφίστε. Πέρα στις φοφορίες. εγκρίθηκε με τεράστια διαφορά. 93 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 94 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 95 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 96 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 97 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 98 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 99 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 100 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Να ελέγξουμε. Όχι. 101 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 102-103 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. Συμβιβαστική 4 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 109 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 110 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 111 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 112 υπέρ, κατά,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 128 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 129 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 130 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 131 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 132 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 134 υπέρ, Α, είναι ίδια, λέει ο πρόεδρος. Ποια έχει αποσυρθεί? Καλώς. 135 τότε υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 136 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 137 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 138-139 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνονται. 141 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 142 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 143 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 144 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 145 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 150 τώρα. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 151 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 152 και 153 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. 154 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 155 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. 156 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 157 μέχρι 161 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 162 και 163 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 164 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 165 και 166 υπέρ κατά, αποχές, 167 υπέρ, όχι, έχει αποσυρθεί. 168 επίσης, 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μετρολογικές σκέψει τώρα. 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 6 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 7 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 8 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 10 και 11 υπέρ, κατά, αποχές Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά. 10 και 11 ψηφίστε παρακαλώ. Δύο δεν έχουν ψηφίσει. Κοιμούνται, λέει ο πρόεδρος. Πέρα στις ψηφοφορίες εγκρίθηκαν. Η 12 υπέρ, λέει ο πρόεδρος. Α, όχι, καταπίπτει. Έχει εγκριθεί ουσιαστικά. Ναι. 13 τώρα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 14 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 15 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 16 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 17 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 18 και 19 συν προφορική 2, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές θα ελέγξουμε.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 αποχές εγκρίθηκε. 30. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 34 υπέρ, λέει ο πρόεδρος. Α, ξέχασατε 2. 2 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τριάντα τώρα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα της προφορίας Απορρίφθηκε. Δεύτερο τμήμα καταπίπτει, συνεπώς. 40 τώρα. Το κύριου Επιτίδιου υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 41 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 42, 43, 44 και 45. Όχι, 44 έχει αποσυρθεί. Οι υπόλοιπε υπέρ, κατά αποχές απορρίπτονται. 46 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτονται. 47 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτονται. 48 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτονται. Συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 50 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 51 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία τώρα, επί της τροποποιημένης γνωμοδότησης. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Ένα συνάδελφο δεν έχει ψηφίσει ακόμα. Α, τώρα εντάξει, έχουμε ψηφίσει όλοι. Εγκρίθηκε 47 υπέρ 9 κατά συγχαρητήρια. Παρακαλώ κύριε Παντζέρη. Τώρα που ψηφίσαμε, παρακαλώ τον Πρόεδρο να κάνει μια επαλήθευση, γιατί δεν υπάρχουν κανόνες σε σχέση με την ε, επαφέ ανάμεσα στην ΑΦΕΤ και τη ΛΥΜΠΕ. Και υπήρξε ένα αυθαίρετο κριτήριο για το να καθορίσουμε αν μια τροπολογία θα πρέπει να ψηφιστεί εδώ ή αν είναι αρμοδιότητα της ΛΥΜΠΕ. Ε, και κάποιες λογικές τροπολογίες τις οποίες ε, συμμεριζόταν και η συγχύτρια. Γι' αυτό πιστεύω πως είπαμε όχι σε πολύ σημαντικές τροπολογίες που εάν είχαν υπερψηφιστεί θα είχαν ενισχύσει αυτή την έκθεση στην Επιτροπή ε, ΛΥΜΠΕ. Ίσως λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει και μια ρυθμιστική επαλήθευση σε σχέση με τις αρμοδιότητες γιατί φορτικά θα κάνουμε μόνο πολιτικά βάχαλα. Ευχαριστώ κύριε Παντζέρη. Άλλος. όπως σας πρότεινα, νομίζω πως θα πρέπει να συζητήσουμε ε, σε αυτήν την ε, περίπτωση για το πώς θα πρέπει να προχωρήσουμε στο μέλλον ε, για τις εκθέσεις όπου μια επιτροπή δίνει την γνωμοδότησή της και μετά ψηφίζει τις τροπολογίε. Τι είπατε ακριβώς, ε, από ό,τι κατάλαβα δεν είμαστε ικανοποιημένοι, ε, ούτε κι εγώ είμαι ικανοποιημένο με αυτή ε, τη διαδικασία, αλλά αυτή την λύση βρήκαμε και κύριε Παντζέρ θα το συζητήσουμε στο επόμενο διευρυμένο Προεδρείο. Ωραία, σας ευχαριστώ και περνάμε στο επόμενο σημείο, το υπαριθμό 9, ανιθαγένεια στην Νότια και Νοτιοανατολική Ασία. Εισηγητή είναι ο κύριο Μπασίρ. Θέλετε να πείτε κάτι? Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για την εξαιρετική φύση της συνεργασίας μας. Αυτό μόνο. Ευχαριστώ πολύ. Wonderful. Υπέροχα. Μπορούμε να ξεκινήσουμε την διαδικασία ψηφοφορίας, λοιπόν. Ε, τροπολογία 74. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 73. Υπέρ. Ε, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 76 ε, πρέντα. Υπέρκατα. κατά αποχές Α, μάλιστα, ε, πλειοψηφία. 78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 79. Εδώ έχουμε ψήφο με προφορική ε, τροπολογία 1. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 81. Ψευπροφορική τροπολογία 2. Το εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 82 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 84 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 85 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 86 υπέρ κα, κατά, υπέρ μάλλον κατά Α, συγγνώμη, διορθώνει ο πρόεδρος, 88 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 86 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 87 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 89 υπέρ κατά αποχές. Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την 89, για να ξυπνήσουμε λίγο όλοι. Three, two, two colleagues still sleeping. Okay. Δύο ακόμη ψηφίστε. Πέρας. Oh, myself, I was sleeping. Yeah. No, I did vote. No, Όχι, ψήφισα εγώ. Oh, okay. But it's been carried with 36 to 21. Ναι, εντάξει, εγκρίθηκε 36 κόντρα 21. Λοιπόν, τροπολογία 90. That was a good one. Uh, amendment 90 in favor. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύε 1, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύε 2, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 91 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 92 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 93 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 94 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 95 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 96 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 97 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 98 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 100 υπέρ κατά αποχές αυτό έπρεπε να έχει απορριφθεί. Απορρίφθηκε. 99 επέρ, Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Φτάνουμε στην 102 και την 103 υπέρ υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Ε, το 104 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. 105 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 107 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 106 υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται. 108 υπέρ. Έλα παιδιά, τα χέρια ψηλά. 108 υπέρ κατά. Εγκρίνεται σίγουρα. 109 υπέρ κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 110-111 υπέρ κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 112 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 113 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 114-115 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 116 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 117 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 118-119 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 120 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 121 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 122 υπέρ κατά αποχές κατά απορρίπτεται 123 ε, υπέρ κατά αποχές εκείνεται 124 υπέρ κατά αποχές εκείνεται 125 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται μου φαίνεται έλεγχος ηλεκτρονικός εντάξει 125 ελέγχουμε ηλεκτρονικά Δύο λοιπόν πέρασε. 21 υπέρ, 36 κατά απορρίπτεται. Πάμε τώρα στην 126. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εξαιρετική υπερψήφιση. 127 ε, και 128. Ε, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. Τροπολογία 130 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 129 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πάμε στην ΔΕΒΕ 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. ΔΕΒΕ 4 υπέρ κατά αποχές εγκρινεται ΔΕΒΕ DV5 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε ΔΕΒΕ DV5 άρχεται η ψηφοφορία. The vote is closed. That has been carried. Εγκρίνεται. Ε, 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 136 και 137, Σαφχάουζερ Πρέντα. Είναι ταυτόσιμες. Remarkable, in favor. Τι να πει κανείς. Υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Ναι. Εγκρίνεται. Εγκρίνονται. εγκρίνηθηκαν. Ε, ΔΕΒΕ 8 υπέρ κατά αποχές. Σήκωσε κανείς χέρι. Όχι. Ξανά. ΔΕΒΕ 8 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. ΔΕΒΕ 7 ε, υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. απορρίπτεται. Συγγνώμη. Τροπολογία 12. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 13. Υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στην ΔΒΒ. Voted on compromise 5. Uh, where do we go now? DVB. Where's DVB? Oh, over there. Next page. DVB. DVB. Τμήμα 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 34 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 36 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. Περνάμε τώρα στην ε, ΔΕΒΕΣΥ. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ερχόμαστε στην 45 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. 46 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. 47 υπέρ κατά αποχές. Να ελέγξουμε αυτήν ηλεκτρονικά τη 47 Τζαμπάσκι. Άρχεται η ψηφοφορία. Κα, ε, τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. 48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 58. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. 58 λοιπόν. Άρχεται. Και τέλος της ψηφοφορίας και απορρίφθηκε. Συμβαστική 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε στην 68. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. 68. Εγκρίνεται υπέρ 70 ε, ε, <coughs> υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 69 α συγγνώμη έχει καταπέσει 71 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 72 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τώρα, τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ κατά αποχές έγκρινται, 5 υπέρ κατά αποχές έγκρινται, 6 υπέρ κατά αποχές έγκρινται, 7 υπέρ κατά αποχές έγκρινται. τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές έγκρινται, τροπολογία 9 υπέρ κατά ελέγχουμε την 9 Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. 30 προς 28. Ε, τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα πρέπει και πάλι να ελέγξουμε. 10 λοιπόν. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Λοιπόν, η... συνάδελφος... Λοιπόν, 30 προς 29, πέρασε. Πάμε στην 11, υπέρ. Κατά αποχές, έλεγχος ηλεκτρονικός και πάλι για την 11. Vote is closed. Uh, 36 to 22. Τέλος ψηφοφορίας, 36 προς 22 εγκρίθηκε. Ψηφίζουμε τώρα ηλεκτρονικά για το σχέδιο ψηφίσματος, όπως τροποποιήθηκε. Άρχεται. Two colleagues missing. Δύο συνάδελφοι λοιπόν δεν ψήφισαν. Πέρασε. 54 ψήφοι προς 2. Συγχαρητήρια ε, στον εισηγητή. Περνάμε στο σημείο τώρα υπερθμών 10. δημοσιονομικοί κανόνες εφαρμόζονται στο Γενικό Προπολογισμό τη Ένωση. Η συγγετή είναι Άντι Χριστέα. Θέλετε να πείτε κάτι. Θέλω να ευχαριστήσω τους εισηγητές, του σκιώδες δηλαδή και τη γραμματεία για την πολύτιμη βοήθειά τη. Ευχαριστούμε. Να αρχίσουμε την ψηφοφορία λοιπόν. Συμβεβαστική ένα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 33 με προφορική ε, τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Περνάμε στην τροπολογία 39. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε αυτήν την 39. Πέρας. Σαράντα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 51 υπέρ τι, για την 50 να ελέγξουμε, εντάξει. 50 έλεγχος Τέλος. Εγκρίθηκε. Λοιπόν, πού ήμασταν. Πάμε στην 51. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Εγκρίνεται. ναι, υπέρ, κατά, αποχές, έγκρινεται. Συμβαστική 3 υπέρ, κατά, αποχές, έγκρινεται. Περνάμε στην τροπολογία 14. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 15 υπέρ, κατά, αποχές, ε, Έλεγχος. «28 προς 26 γίνεται 16 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, ε, γίνεται 16 υπέρ. Τέλος ε, της ψηφοφορίας απορρίφθηκε 16. 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 υπέρ κατά αποχές ε, <clears throat> αποχές έλεγχος ηλεκτρονικός 20 ε, άρχεται, τέλος. Μα τι είναι, χάλα στο μηχάνημα. Όχι, όχι, πάνω από δύο ψήφισαν κατά με τα χέρια πάντως. Βάση περιπτώσει, προχωράμε. Πού ήμασταν στην 21. Ψηφίζουμε. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 22 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 23 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 24 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 25 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία άρχεται. Πέρας. 42 προς 1. Σημείο 11. Έχουμε τη Συμφωνία Σταθεροποίηση και Σύνδεση μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών του, αφενό και τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, αφετέρου, στην ληφθεί υπόψη προσχώρηση τη Δημοκρατία τη Κροατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο μία ψηφοφορία είναι, άρχεται. Μία, μία ψηφοφορία άρχεται. ενα συνάδελφο λείπει. 57 προς 1. Συγχαρητήρια. Right, to Moldova, item number 12. Πάμε τώρα στη Μολδαβία, το σημείο 12, μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στη δημοκρατία της Μολδαβίας. Δεν είναι εδώ η Θέλει κάποιος να πει κάτι άλλο. Όχι, τότε ξεκινά η ψηφοφορία. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 5 υπέρ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 49 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 50 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 52 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 51 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 53 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Να ελέγξουμε. Ωραία. 53. Άρχεται η ψηφοφορία. It's closed. Πέρασε της ψηφοφορίας. 40 προς 17. 54 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 55 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 56 υπέρ, κατά, αποχές, ε, απορρίπτεται. Να ελέγξουμε. Ωραία, 56. Ελέγχουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Είμαστε στο 56, κύριε Σόλτ. Πέρα της ψηφοφορίας. 30 προς 27. Εγκρίνεται. Τώρα έχουμε την 57 έως την 60. Τέσσερις φορές Σαφχάουζερ. Να το κάνουμε όλα μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Όλες απορρίπτονται. 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 61 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 62 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 63. 64. 63 υπέρ αποχές απορρίπτεται, 64 υπέρ αποχές αποχή, 65 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 66 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Πάμε στις αιτιολογικές σκέψεις. 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται.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 Ορίστε, είπατε κάτι. Ποιο. 12. Έχουμε φτάσει στο 15. Το 15. Για να το ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 15. πέρα τη ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Πάμε στη 16 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται έτσι. Να ελέγξουμε. 16 Μανέσκου άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 30 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε. Η 30 καστάντου. Πέρας. Απορρίπτεται. 31. Κύριε Σόλτς, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απο... Εγκρίνεται. 32. Με την προφορική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τελική ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία για το σύνολο της γνωμοδότησης. Ψήφισαν και οι 59 πέρα της ψηφοφορίας, 55 ψήφοι υπέρ, 4 κατά, συγχαρητήρια στον εισηγητή. Ωραία. Θα συνεχίσουμε σε δύο λεπτά τη συνεδρίασή μας. Right, ladies and gentlemen, it's 10 o'clock. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι 10 η ώρα. Συνεχίζουμε τη συνεδρίασή μας και σας παρακαλώ όλους να καθίσετε. Καθίστε όλοι παρακαλώ. Λοιπόν, περνάμε στο σημείο 13 της ημερήσιας διάταξης. Πρόκειται για την ε, συζήτηση όσον αφορά την Βοσνία και Ερζεγοβίνη και με ιδιαίτερη χαρά ε, υποδέχομαι εδώ τον Υπουργό Εξωτερικών της χώρας, τον κύριο Ίγκορ Κντάκ. Εκ μέρους λοιπόν ε, της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων σας καλωσορίζω εδώ. Τον συνοδεύει ο πρέσβης της χώρας, ο κύριος Τόπριτς, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τον έχουμε συναντήσει πολλέ φορέ γιατί συχνά είναι στην ε, ημερήσια διάταξη τη Επιτροπή μα το θέμα της Βοσνίας Ζεγοβίνη. Μια χώρα 25 ετών. Εδώ και δύο χρόνια υπάρχει και ισχύει η συμφωνία που έχουμε με την χώρα αυτή εν ώψη της ε, αίτηση ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι προοπτικέ είναι ιστορική σημασία. Η χώρα σα είναι για μας ε, μια δοκιμή κατά κάποιο τρόπο για το τι συμβαίνει στα Βαλκάνια. Αν εσείς ξεπεράσετε ε, τις προκλήσεις όσον αφορά την ε, ειρήνη και την ε, ανάπτυξη, αυτό θα είναι δείγμα για ολόκληρα τα Βαλκάνια. Τα Δυτικά Βαλκάνια και ιδιαίτερα η Βοσνία, η Ριζεγοβίνη, πέρασε δύσκολες στιγμές τελευταία και κατά το παρελθόν Έχουμε φέτος, εμείς την επέτειο, 60 ετών από την υπογραφή της Εθήκης της Ρώμης, που οδήγησε την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει τη μεγαλύτερη περίοδο ειρήνης ε, ποτέ και πουθενά. Παρόλα αυτά, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έχουμε να θυμόμαστε και αυτά που συνέβησαν στην Βοσνία Ερζεγοβίνη πριν από 22 χρόνια. Κάτι το οποίο είναι βέβαια ιδιαίτερα σοβαρό και τραγικό. Τη σφαγή της Εμπρέβνητσα δηλαδή. Πρέπει λοιπόν να ενισχυθούν οι θεσμοί στο Σαράγεβο και να αποφύγουμε την πόλωση. Να συντονιστούμε για να δώσουμε απαντήσεις, να αποφευθεί το οργανωμένο έγκλημα και η νομοποίηση παράνομου χρήματος. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας ζητήσω να πάρετε το λόγο εδώ μπροστά στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και να μας μιλήσετε για τις προκλήσεις αυτές που αντιμετωπίζει η χώρα σας. Για άλλη μια φορά σας καλωσορίζουμε εδώ μεταξύ φίλων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μακάλιστερ, ευχαριστώ και εσάς και ευχαριστώ επίσης και όλους τους συναδέλφους. Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι ενώπιόν σας για να ανταλλάξουμε απόψεις όσον αφορά την κατάσταση στη Βοσνία Ζεγοβίνη και τις διαδικασίες εκεί. Επιτρέψτε μου να αρχίσω με κάποια σχόλια και μετά θα περάσουμε βέβαια στο πιο ενδιαφέρον θέμα που είναι η συζήτηση των θεμάτων αυτών μεταξύ μας, η ανταλλαγή απόψεων δηλαδή μεταξύ μας. Πρώτα απ' όλα, η Βοσνία Ζεγοβίνα είναι μια χώρα η οποία έχει δεσμευτεί με ιδιαίτερη αποφασιστικότητα προκειμένου να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη Βοσνία Ζεγοβίνη δεν έχουμε πολλά θέματα πάνω στα οποία να συμφωνούμε στην ε, Ομοσπονδία με την ε, Σέρψκα αλλά όλοι συμφωνούμε πάνω σε αυτό. Όλοι θέλουμε η διαδικασία αυτή ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχιστεί και να πετύχει όσο γίνεται πιο γρήγορα και όσο γίνεται πιο αποτελεσματικά. Μία από τις τελευταίες έρευνες δείχνει ότι πάνω από 80% του πληθυσμού της χώρας στηρίζει τη διαδικασία αυτή προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να γίνει δηλαδή η Βοσνία Ζεγοβίνη μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Βοσνία Ζεγοβίνη όσον αφορά την εξωτερική της πολιτική Δύο ζητήματα κυριαρχούν και έχουν προτεραιότητα για μας. Η διαδικασία ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το ένα και η περιφερειακή συνεργασία είναι το δεύτερο. Και τα δύο αυτά είναι πράγματα τα οποία μας βάζουν στον δρόμο αυτό προς την ένταξη. Θα σας μιλήσω και για τα δύο. Πρώτον, το 2016 ήταν η χρονιά των μεγαλύτερων αλλαγών και της μεγαλύτερης προόδου που έχει επιτευχθεί ποτέ στη χώρα στον δρόμο αυτό της ένταξης. Τέτοια πρόοδο δεν είχαμε κάνει καμία άλλη χρονιά. Και αυτό έγινε, το πετύχαμε και χρονιά εκλογών που είχαμε στη Βοσνία Ζεγοβίνη, κάτι που όπως καταλαβαίνετε καθιστά ακόμα πιο σημαντική την πρόοδο αυτή. Αυτό που χρειαζόμαστε τώρα δεν είναι να σταματήσουμε, αντίθετα είναι να έχουμε μια επίσης πολύ καλή χρονιά το 2017. Ξέρετε ότι το ερωτηματολόγιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάρχει από το Δεκέμβριο στη χώρα και είναι στα ευρωπαϊκά ζητήματα που επικεντρώνουμε περισσότερο την προσοχή μας. Πρόθεσή μας και επιθυμία μας είναι να γίνουμε υποψήφια χώρα όσο γίνεται πιο γρήγορα ή δυνατόν πριν το τέλος της χρονιάς αυτής. Και θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται προκειμένου να το πετύχουμε. Η διαδικασία ένταξης της Βοσνίας Αρζεγοβίνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ελπίζω και συνάδελφοι από τα Δυτικά Βαλκάνια ή άλλες ε, χώρες που οι υποψήφιες να μην ε, διαφωνήσουν, η διαδικασία ένταξης της χώρας μου στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τη μεγαλύτερη δυνατόν σημασία. Μπορεί για μας μάλιστα να είναι ακόμα μεγαλύτερη σημασία από ό,τι είναι για άλλες χώρες. Γιατί η ειρήνη, η σταθερότητα διαρκείας και μια συμφωνία διαρκείας μεταξύ όλων εμάς που βρισκόμαστε στη Βοσνία Ζεγοβίνη είναι κάτι εφικτό μόνο εφόσον υπάρχει αυτή η ευρωπαϊκή προοπτική. Και αυτό μπορεί να πετύχει μόνο εφόσον είναι ορατό το σημείο ένταξης τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν μιλήσετε με οποιονδήποτε στην Βοσνέζο, είτε στη Μόστρα, είτε στη Πανιαλούκα, είτε στο Σαράγεβο, θα δείτε ότι όλοι το θέλουν Και υπάρχουν τρία στοιχεία εδώ. Το ένα είναι ότι θα υπάρξει οικονομική πρόοδος, ότι δεν θα έχουμε πια, για παράδειγμα, 60% ανεργία μεταξύ των νέων. Αυτό θα σταματήσει. Και είναι σαφές γιατί οι νέοι, άντρες και οι γυναίκες θέλουν να φύγουν από τη χώρα. Υπάρχουν οικονομικοί λόγοι. Όμως, ο κόσμος στη χώρα βλέπει τη διαδικασία αυτή σαν μια εξασφάλιση επιτυχίας του κράτους δικαίου. Γιατί ο κόσμος παραπάνω και από την δουλειά και την οικονομική ανάπτυξη αυτό που θέλουν είναι δικαιοσύνη. Θέλουν δικαιοσύνη, θέλουν κράτος δικαίου, το οποίο είναι εξίσου σημαντικό όπως και η οικονομική ανάπτυξη. Συνεπώς, το βλέπουν σαν εξασφάλιση αυτό, αυτή την πορεία οι κάτοικοι της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Οι περισσότεροι πολίτες έχουν ζήσει ένα, δύο, ακόμα και τρεις πολέμους. Αν λοιπόν η διαδικασία ένταξης και η ολοκλήρωση στην περιοχή σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν πια πόλεμοι, ακόμα και αν δεν υπήρχε κανένα άλλο όφελος δηλαδή, αλλά μόνο το ότι δεν θα υπάρχουν πια πόλεμοι για τα επόμενα 100 χρόνια, αυτό θα έφτανε για μας. Για να σας εξηγήσω πώς ο κόσμος βλέπει αυτή τη διαδικασία πως οι πολίτες ολόκληρη τη Βοσνία Ζεγοβίνη βλέπουν την πορεία αυτή και γιατί θέλουν τόσο πολύ την προσχώρησή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θέλουμε και την περιφερειακή συνεργασία. Έχουμε δεσμευτεί και από αυτού και βλέπουμε τις ευκαιρίες που προσφέρει μια τέτοια περιφερειακή συνεργασία με τους φίλους μας στη Σερβία, το Μαυροβούνι, την Μακεδονία και άλλες, περιοχές, και άλλες χώρες στην περιοχή. Πιστεύουμε ότι είναι πλεονέκτημα για μας να έχουμε τα μεγαλύτερα σύνορα με την Κροατία που είναι πάνω από 1000 χιλιόμετρα που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκείνη και για μας είναι και αυτό μια ευκαιρία για να επιταχύνουμε τη διαδικασία ένταξής μας. Ποια είναι τώρα τα εμπόδια. Είναι σημαντικό εδώ να πούμε ότι το πιο γενικό αλλά και το πιο επικίνδυνο εμπόδιο είναι το θέμα της πολιτικής σταθερότητας στη χώρα. Στη Βοσνία Ζεγοβίνη, όπως γνωρίζετε, έχουμε τη συμφωνία ε, του Ντάλτον. Ξέρετε ότι αυτή αποτελεί την ε, βασική μας, ε, το βασικό μας στοιχείο και αυτό το οποίο θέλουμε είναι να συνεργαστούμε μεταξύ μας, να έχουμε αμοιβαία κατανόηση, να έχουμε διάλογο μεταξύ μας και είναι ο μόνος τρόπος για να πετύχουμε. Ο καθένας έχει τις δικές του απόψεις. Αν μιλήσετε ε, με τον κόσμο στα διάφορα σημεία της χώρας, εκπροσώπους δηλαδή των ε, διαφόρων ε, περιοχών, θα ακούσετε διαφορετικές απόψεις όσον αφορά το παρελθόν. Αλλά γι' αυτό και λέμε ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στο μέλλον και να καθίσουμε και να συζητήσουμε και να βρούμε κοινό τόπο για τη μελλοντική μας πορεία. Είμαστε μπροστά στα επόμενα βήματα όταν μιλάμε για την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι λοιπόν σημαντικό να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις. Έχουμε ένα θεματολόγιο για μεταρρυθμίσεις που εκπονήσαμε από κοινού με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πέρασε, εγκρίθηκε κάτι το οποίο δεν συμβαίνει συχνά στη Βοσνία Ζεγοβίνη. εγκρίθηκε ομόφωνα από όλους. Ακόμα και από την αντιπολίτευση, τα κόμματα της αντιπολίτευσης συμφώνησαν και οι δικοί τους βουλευτές συμφώνησαν. Και η δήλωση αυτή υπογράφηκε από όλους τους επικεφαλείς των ε, πολιτικών κομμάτων, ακόμα και αυτών που βρίσκονται στην αντιπολίτευση. Συνεπώς συνεχίζουμε και επικεντρωνόμαστε περισσότερο στα οικονομικά ζητήματα, τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις, και αυτές είναι οι κυρίες προσπάθειές μας αυτή την εποχή. Η Βοσνία Ερζεγοβίνη τώρα, όσον αφορά τις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν μιλήσουμε θεσμικά, έχουμε το ζήτημα της κοινοβουλευτικής συνεργασίας. Αυτό το ζήτημα λοιπόν, το κοινοβουλευτικό, οι σχέσεις της Βοσνίας Ερζεγοβίνης με την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σταματήσει κάπως. Μίλησα με κάποιους ευρωβουλευτές και ελπίζω ότι θα μπορέσει να λυθεί. Οι διάφορες διαδικασίες δηλαδή που πρέπει να αναλυθούν για να προχωρήσουμε σε αυτό. Όπως είπα και στην αρχή, είναι ενδιαφέρον να ανταλλάξουμε και απόψεις μεταξύ μας και να ακούσω βέβαια και τις δικές σας απόψεις, τι λέτε για την Κοσνία ε, Αρζακοβίνη και την διαδικασία ενταξής μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ για τις αγωγές σας αυτές τις παρατηρήσεις. Έχουμε 40 λεπτά για όλο αυτό το θέμα. Έχω 12 συναδέλφους που έχουν ζητήσει το λόγο, οπότε παρακαλώ μένετε στα δύο λεπτά έκαστος και θα ξεκινήσουμε με τον πρόεδρο της ε, αντιπροσωπείας για την Βοσνία και Ζεγοβίνη και το Κωσυφοπαίδιο, τον κύριο Πίτσουλα. Σας ευχαριστώ. Είναι μεγάλη μας χαρά πραγματικά να έχουμε σήμερα μεταξύ μας τον Υπουργό των Εξωτερικών Υποθέσεων της Βοσνίας Ριζεκοβίνης, τον, Ήβο, τον κύριο Ήβο Τσαρνάκ. Ε, δείχνει αυτό πόσο πολύ είναι προσδεδεμένος, αφοσιωμένος στην ε, ε, ευρωπαϊκή πορεία της χώρας του και είναι πάρα πολύ καλό που μας θύμισε όλες τις επιτυχίες που σημειώθηκαν το 2016 στη χώρα του ε, ε, παρά τα εμπόδια που ορθώθηκαν σε αυτή την πορεία. Μας δείχνει ότι είναι δυνατόν να προχωρήσει η χώρα αυτή παρά τις δυσκολίες και παρά τα διορθωτικά προβλήματα. Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να επανέλθω σε ένα πρόβλημα, μία δυσκολία που πιστεύω πως ε, αυτό είναι που ενοχλεί τις σχέσεις με μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη Βοσνίας Ζεζεγοβίνη. Ε, πρόκειται για τι σχέσει ανάμεσα στα κοινοβούλια. Εμείς ε, δεν υπάρχει αφιβολία γι' αυτό. Θέλουμε η Βοσνία Ζεγοβίνη να ευημερήσει και να σταθεροποιηθεί, αλλά φυσικά πρέπει πρώτα απ' όλα να λειτουργήσει ω κράτο και η προσχώρηση στο Ευρωπαϊκό, ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο με συνένεση. Δυστυχώ, οι σχέσεις, μάλλον μέσα στι σχέσει ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Βοσνία Ζεγοβίνη, η κοινοβουλευτική διάσταση δεν υπάρχει. Δεν έχει συσταθεί μειχτή επιτροπή σύνδεσης και σταθεροποίησης έχουμε προσκρούσει σε ένα τεχνικό και πολιτικό πρόβλημα σημαντικό και για την ώρα δεν φαίνεται να υπάρχει λύση παρά τις απόπειρες. Φαίνεται πως το κοινοβούλιο της χώρας φοβάται πως θα χάσει κάποιες προϋποθέσεις, κάποιους όρους που εγγυώνται την ε, θέση του. Πώς μπορείτε εσείς να συμμετέχετε σε αυτή τη διαδικασία, εφόσον δεν είμαστε σε εκλογικό έτος, πώς μπορούμε να προσπαθήσουμε να φέρουμε πιο κοντά τις θέσεις μας και να βοηθήσουμε την Βοσνία Ζεγοβίνη να έρθει πιο κοντά στην Ένωση, πράγμα που επιθυμούμε φυσικά όλοι μας. Ε, ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πρέντα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ κύριε Υπουργέ που είστε εδώ ώστε να μιλήσουμε για μεταρρυθμίσεις που έχει κάνει η χώρα. Σας ευχαριστώ που είστε σήμερα εδώ λοιπόν για να μιλήσουμε για αυτές τις μεταρρυθμίσεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια. Ε, συμφωνώ μαζί σας όταν λέτε πως είναι μια περίοδος προόδου, ειδικά αν δούμε τι συνέβαινε στο παρελθόν και συγκρίνουμε. Ε, έχω τρεις ερωτήσεις αν μου επιτρέπετε. Η πρώτη αφορά την συζήτηση όσον αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για τα καύσιμα και τα προϊόντα πετρελαίου. Είναι πολύ σημαντικό φόρος αυτό για να μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν διάφορα μέτρα. Προβλέπεται εξάλλου και στην ατζέντα για τη μεταρρύθμιση και όλες οι, χώρες, οι δυνάμεις της χώρας συμφώνησαν σε αυτό. Ποιες είναι οι πιθανότητες να εγκριθεί εγκαίρως αυτή η νομοθεσία, γιατί βλέπουμε να ε, υπάρχει μεγάλη ένταση. Δεύτερον, προετοιμασία των απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο. Πότε θα γίνει αυτό. Ε, είδαμε να επικρατεί η αισιοδοξία στην αρχή, αλλά τώρα έχω την εντύπωση πως έχουμε λίγο φρενάρι. Και τελευταία ερώτηση, είδαμε τη δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε πρόσφατα από την ΑΕΡΑΕ ε, όπου διαπιστώνεται μια σημαντική διαφορά ανάμεσα στην στήριξη υπέρ της ένταξης ε, της ε, Ένωσης στη Ρεπούμπλικα Σέρβσκα. Εσείς είστε από την Ρεπούμπλικα Σέρβσκα. Τι μπορούμε να κάνουμε εκεί για να αλλάξει κάπως γενικώ η στάση, γιατί δεν είναι μόνο Ντόντικ η Ρεπούμπλικα Σέρβσκα. Τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε τους όσους είναι υπέρ της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Ε, Σκιώδης. Ο κύριος Παπαδάκης. Να καλωσορίσουμε τον Υπουργό Εξωτερικών της Βοσνίας Αζεγοβίνης. Να του πω ότι πρόσφατα ανέλεβα σκιώδης εισηγητής εκ μέρους της ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Προέρχομαι από την Κύπρο, η οποία και αυτή έχει σοβαρότατα προβλήματα και μπορώ να αντιληφθώ σε πολύ μεγάλο βαθμό τις δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζετε. Δύο-τρία σημεία θέλω να δείξω πολύ γρήγορα. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό για να υπάρξει προοπτική, ιδιαίτερα προς τις νέες γενιές, είναι να κυλήσουν γρηγορότερα μεταρρυθμίσεις, ούτω ώστε να νιώθουν ότι κάτι αλλάζει στη ζωή τους. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό σημείο είναι η καταπολέμηση της διαφθοράς, η οποία καθημερινά απογοητεύει τους νέους και τους αποστρέφει από την υπάρχουσα εγκατάσταση με αποτέλεσμα να θέλουν να φύγουν από τη χώρα. Και το τρίτο σημαντικό είναι τι ρόλο παίζουν οι θρησκευτικοί ηγέτες στη χώρα σας. Γιατί θεωρώ εάν λειτουργήσουν με έναν τρόπο ούτω ώστε να αμβληθούν οι διαφορές τα πράγματα θα είναι πολύ πιο εύκολα και καταλαβαίνουμε όλοι τι συμβαίνει σήμερα με την όξυση των θρησκευτικών διαφορών θα πρέπει να υπάρξει πίεση προς αυτήν την κατεύθυνση ούτως ώστε να υπάρξει εξομάλυση των σχέσεων και να λειτουργήσουν ως ενοποιητικό στοιχείο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. And now we come to Mr. Ευχαριστώ κύριο Στάνοκ, εκ μέρους του ECR. Ευχαριστώ Πρόεδρε, φυσικά η ομάδα μου υποστηρίζει την υποψηφιότητα της Φωσνίας Ερζεγοβίνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, όχι όπως το Κόσοβο, επειδή δεν το έχουμε αναγνωρίσει. Είναι άλλη μία χώρα η οποία θέλει να γίνει υποψήφια όμως ε, μας δείχνει και τη δουλειά που πρέπει να γίνει. Ο, ρόλος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης είναι ακόμα αδύναμος και υπάρχουν φυγόκεντρες ε, δυνάμεις που επηρεάζονται και από την ανάμειξη της Ρωσίας ε, στην περιοχή. Εδώ και μια δεκαετία από τότε που έγινε η συμφωνία του Dayton. Ε, έχουμε πολλές προκλήσεις ακόμα. Έχουμε παρόλα αυτά στην ομάδα μας κάθε μορφής υποστήριξη προς ε, την υποψηφιότητα και θέλουμε να βοηθήσουμε τη χώρα για την προσχώρησή της. Δύο ερωτήσεις. Ποιος είναι ο ρόλος της Ρωσίας. Φυσικά είναι γνωστός. Εγώ είμαι ο εισηγητής για το Μαυροβούνιο και έχουμε δει τις δραστηριότητες εκεί. Θέλουμε όμως να, να ξέρουμε και ποιος είναι ο ρόλος της Τουρκίας στη χώρα σας και ειδικότερα ένα σχετιζόμενο ερώτημα είναι ε, πώς γίνεται εξωτερική χρηματοδότηση των ε, φιλανθρωπικών οργανώσεων, των ε, τζαμιών ε, των σαλαφιστών, τι γίνεται με τους ε, τζιχαντιστές που έχουν φύγει από τη χώρα σας και μπορεί να επιστρέψουν με την επερχόμενη ήττα του ISIS στη Ράφα και θέλουμε να μάθουμε και κάτι άλλο που έχει να κάνει με το ρόλο του Ηνωμένου Βασιλείου μετά το Brexit. Μου είπαν ότι η εξωτερική υπηρεσία εξωτερικής δράσης ε, δεν θέλει η Σύνοδος Κορυφής ε, για την ατζέντα του Βερολίνου να γίνει του χρόνου στο Λονδίνο λόγω του Brexit. Εσείς ε, τι πιστεύετε για την Μεγάλη Βρετανία, πρέπει να μείνει στο πεδίο και μετά τον Brexit. Ευχαριστούμε τον Τσάρλς, ο κύριος Ράτος για τους ε, φιλελεύθερους. Ευχαριστώ Πρόεδρε, σας, ε, κύριε Υπουργέ, σας εύχομαι κάθε υποστήριξη από την ομάδα μου ε, για την ε, Βοσνία το στο δρόμο της ε, προς την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν από λίγο εγκρίναμε ένα πρωτόκολλο για τη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης που έχει να κάνει και με την προσχώρηση της Κροατίας. Προχωρούμε και εκεί υπάρχουν και άλλες συνθήκες και όροι όπως είναι η εφαρμογή του σχεδίου μεταρρυθμίσεων και του μηχανισμού συντονισμού για να μπορέσει να προχωρήσει μια τέτοια διαδικασία. Η Εκτελεστική Επιτροπή, λοιπόν, ε, πρέπει να μας δώσει τώρα κάποιες απαντήσεις, ε, οι οποίες πρέπει να αντικατοπτρίζουν την πολιτική κατάσταση στη Βοσνία Ριζεγοβίνη. βάση, λοιπόν, του ερωτηματολογίου αυτού, θα ξεκινήσει και πάλι μια διαδικασία για το μηχανισμό συντονισμού ε, και θα είναι και ένα τεστ ε, για το μέλλον, γιατί οι μηχανισμοί αυτοί είναι πραγματικά κάτι πολύπλοκο, τα πιο πολύπλοκο πράγμα που έχουμε δει για μια χώρα ε, υπό ένταξη. Πώς λειτουργεί λοιπόν αυτός ο μηχανισμός μέσα στα πλαίσια των ερωτήσεων που έχουν να κάνουν και με το ερωτηματολόγιο που έχουμε δώσει στην Εκτελεστική Επιτροπή. Ωραία. Ευχαριστούμε συνάδελφοι. Ένας πρώτος γύρος ομιλητών με τόσες ερωτήσεις. Πρέπει λοιπόν ο Υπουργός Εξωτερικών να απαντήσει πρώτα στον πρώτο γύρο και μετά αν έχουμε χρόνο θα κάνουμε και ένα δεύτερο γύρο. Πριν απαντήσετε κύριε Υπουργέ να σας ρωτήσω, υποστηρίζετε την ιδέα της Τελωνιακής Ένωσης των Δυτικών Βαλκανίων και τι πιστεύετε μπορούμε να κάνουμε μια ε, ε συνοδοκορυφή για το θέμα αυτό στην Τεριέστη. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις ε, σε αυτό το πρώτο γύρο. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος για να έχουμε και άλλες ερωτήσεις. Καταρχώς ε, για τον κύριο Πίτσουλα για το μεικτό κοινοβουλευτικό συμβούλιο. Τι μπορεί να γίνει γι' αυτό. Ξέρουμε αυτό το διαχωρισμό μεταξύ της ε, κυβέρνησης, στη δική μας περίπτωση, δηλαδή το Συμβούλιο των Υπουργών και του Κοινοβουλίου. Ξέρουμε πόσο ευαίσθητη είναι αυτή η ισορροπία. Πρέπει να πάμε αργά-αργά, αλλά σίγουρα θα έχουμε και συνομιλίε με του ανθρώπους που εκπροσωπούν το κοινοβούλιο μα για να δούμε αν υπάρχει δυνατότητα να προσπαθήσουμε να γίνουμε κομμάτι μια λύση που θα έρθει τις επόμενε εβδομάδες, γιατί τώρα είναι πραγματικά η στιγμή γι' αυτό. Και σίγουρα κατανοούμε το πρόβλημα. Είναι απλώς ένα μείγμα κάποιων εκ των φόβων, ε, κάποιων εκ των πραγμάτων που λαμβάνουν χώρα, εντός της χώρας μας, κάποιες μάχες, κάποιες διαμάχες και τώρα έχουμε την δυνατότητα πλέον να ρυθμίσουμε όλα τα εσωτερικά μας ζητήματα και τις διαδικασίες μέσω της συνεργασίας μας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για μένα λοιπόν είναι αδύνατο να σας δώσω λύσεις αυτό, αυτή τη στιγμή. Ξέρω ότι υπάρχουν κάποιες συστάσεις και θα προσπαθήσω να λάβω μέρος στις συνομιλίες εντός της χώρας για αυτό το θέμα. Τώρα για τις ερωτήσεις που έρχονται από τον κύριο Πρέντα. Ένα από τα πιο ε, καυτά ζητήματα τώρα είναι η η κατάσταση. Οι νέοι νόμοι, ένα πακέτο τεσσάρων νόμων για τα πετρελοειδή και κάποια άλλα είδη φορολογίας. Υπάρχει μια εσωτερική πολιτική μάχη, θα χάσουμε πολύ χρόνο πριν μπούμε στις, για να μπούμε στις λεπτομέρειες, όμως για να καταλάβετε να σας πω ότι έχουμε διάφορα κόμματα που συμμετέχουν στην κυβέρνηση ε, στις διάφορες οντότητες και στο Συμβούλιο των Υπουργών σε κρατικό επίπεδο και υπάρχουν και όροι για το πώς περνούν αυτοί οι νόμοι μετά από τις εσωτερικές πολιτικές διαμάχες, γιατί κάποια από τα πολιτικά κόμματα θέλουν να ε, έχουν υποστήριξη για τους καλλιεργητές που πλήττονται περισσότερο από τους νέους νόμους. Και γι' αυτό θέλουμε όλο το πακέτο να είναι αποδεκτό από όλους. Δεν υπήρξε κάποια λοιπόν τέτοια συμφωνία και δεν πέρασε το, με την διαδικασία του κατεπήγοντος αυτό ε, το θέμα από το Κοινοβούλιο. Δεν ξέρουμε πώς θα προχωρήσει το θέμα. Υπάρχει πιθανότητα να περάσει γρήγορα, αν αλλάξουν οι διαθέσεις. Αλλά κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για το πότε και πώς θα ε, αντιμετωπιστεί αυτό το πακέτο των τεσσάρων ε, νόμων στις επόμενες εβδομάδες και αν θα περάσει γέρος, ειδικότερα για να αντιμετωπίσουμε τις, τα deadlines, τις προθεσμίες του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για να πάρουμε τη δεύτερη δόση από αυτούς. Τώρα, για τις ε, ερωτήσεις που είχαν να κάνουν με το ερωτηματολόγιο. Είναι λίγο πολύ ίδια ερώτηση με αυτή που ανέφερε ο κύριος Ράντος. Μας πηγαίνει στον μηχανισμό συντονισμού. Αυτός ο μηχανισμός είναι όπως ακούσαμε μάλλον ο πιο περίπλοκος μηχανισμός που υπήρξε ποτέ οπουδήποτε. Και ακόμα δεν ξέρουμε πώς θα λειτουργήσει. Έχουμε πάρει μια πολιτική απόφαση για τη δημιουργία του πρόσφατα. Ομόφωνα αποφασίσαμε όχι μόνο σε επίπεδο κράτους αλλά και σε ε, επίπεδο κοινοτήτων. Το θέμα όμως είναι αν θα λειτουργήσει αυτό. έχουμε ακόμα φτιάξει το καλύτερο αυτοκίνητο, αλλά είναι ακόμα στο γκαράζ. Όταν το βγάλουμε στο δρόμο θα δούμε. Γιατί οι θεσμοί δίνουν τις δικές τους απαντήσεις στις ερωτήσεις από το ε, ερωτηματολόγιο της Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σε επίπεδο ομοσπονδία, σε επίπεδο κρατηδίων, ε, Ρεπούμπλικα Σέρψκα και τα λοιπά. Και όλα αυτά είναι ε, ακόμα ε, σε ζήμωση. Ε, στις επόμενες εβδομάδες θα δούμε πώς ε, θα εξελιχθεί πώς θα βελτιώσουμε και θα, την κατάσταση βάσει των απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο και αν λειτουργεί ο μηχανισμός συντονισμού για την Ρεπούμπλικα Σέρψικα και τη γενική διάθεση και στάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν νομίζω ότι είναι αρνητική. Εγώ είμαι από εκείνη και Είμαι αντιπρόεδρος του κόμματος που το 1999 το είχαμε θέσει ως ε, top προτεραιότητα. Ε, στο νούμερο στις πέντε πρώτες προτεραιότητες. Τότε δεν ήταν και πολύ δημοφιλής η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πραγματικά να σας πω ότι μετά από τόσα χρόνια συνεχίζουμε με την ίδια διάθεση. Δεν υπάρχει τίποτα που να θυμίζει αντιευρωπαϊσμό στην Ρεπούμπλικα Σέρψκα. Αντίθετα, εμείς ε, ε, οι άνθρωποι εκεί θεωρούν ότι είναι Ευρωπαίοι, ε, ότι ανήκουν στην Ευρώπη και θέλουν να ακολουθήσουν τον ευρωπαϊκό δρόμο. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν θα μπω σε πολλές λεπτομέρειες λόγω της έλλειψης χρόνου, όμως είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε αυτό το διαχωρισμό μεταξύ της θέλησης ε, και της ε, βούλησης ε, των ανθρώπων να, να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κάποιον στην κυβέρνηση εκεί. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Υπήρξε μία ερώτηση από τον κύριο Παπαδάκη για το ρόλο των διαφόρων θρησκειών και των ηγετών τους στη χώρα. Πολλές φορές στο παρελθόν, ειδικότερα πριν τον πόλεμο, κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά τον πόλεμο, είχαμε προβλήματα. Όμως, εκ μέρους και των τριών βασικών θρησκειών, αλλά και των άλλων, θα μπορούσα να πω ε, ότι έχουμε μια προσέγγιση που είναι πλήρως αποδεκτή και πλήρως επικοδομητική. Θρησκευτικά λοιπόν έχουμε εκπροσώπηση και για το Ισλάμ και για την Καθολική και για την Αρθόδεξη Εκκλησία. Φυσικά υπήρξαν πολλά που υπόθηκαν σχετικά με την επιρροή στην πολιτική σε καθημερινό επίπεδο από τους θρησκευτικού ηγέτες. Εγώ δεν έχω αυτή την εντύπωση. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται όταν κάποιος λαμβάνει αποφάσεις προσωπικά, όμως γενικά εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ μικρή αυτή η επιρροή. Είναι η μικρότερη που θυμάμαι ποτέ και αυτό είναι καλό νομίζω. Γιατί έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα, να υπάρχει και μια διχογνωμία. Ε, τώρα για την κατάσταση με τους ηγέτες του Ισλάμ είναι σημαντικό να πούμε ότι ήταν πολύ ξεκάθαρη ως προς τη μάχη κατά της τρομοκρατίας και του ριζοσπαστικοποίησης. Η Βοσνία Ριζεγοβίνη είναι πολύ αποφασισμένη και δεσμευμένη και αφοσιωμένη στην παγκόσμια συμμαχία. Προσπαθεί να κάνει το καλύτερο. Η υποστήριξη από τους θρησκευτικού ηγέτες σε αυτό είναι πολύ σημαντική. Τώρα για να απαντήσω στις ερωτήσεις του κυρίου Τάνοκ, γιατί και αυτές εντάσσονται σε αυτό, ε, να πω όμως ε, καταρχάς για το ρόλο της Ρωσίας. Ο ρόλος της Ρωσίας στην Βοσνία Ερζεγοβίνη, ειδικά όταν ε, την θεωρούμε έτσι κάπως μυστικιστική και υποχθόνια, νομίζω ότι μάλλον ε, υπερβάλλουμε. Έχουμε συμφέροντα φυσικά ε, ενδιαφέρονται για την Βαλκάνια και την Βοσνία Ερσεγοβίνη. Έχουν και επενδύσεις από όσο ξέρετε σίγουρα στη Ρεπούμπλικα Σέρψκα, αλλά από άποψη πολιτικής επιρροής δεν έχουμε τέτοια επιρροή που να κρούει τον κόδωνα του κινδύνου. Εγώ ως εξωτερικός υπουργό, υπουργός εξωτερικών έχω συναντηθεί με τον κύριο Λαυρόφ ε, πολλές φορές, έχω συναντηθεί Πολλές φορές επίσης και με τον πρέσβη της χώρας έχουμε πάντοτε αποδοχή για τις αποφάσεις μας, που είναι καλές σχέσεις με τη Ρωσία, Έχουμε 5-6 εταιρικέ σχέσεις εξωτερικού εμπορίου, αλλά για μας η στρατηγική στην εξωτερική πολιτική νούμερο ένα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν υπάρχουν λοιπόν εμπόδια ή αρνητικά σχόλια γι' αυτό. Ε, επίσης υπάρχει αυτό το θέμα με, τα φιλανθρωπικά ιδρύματα. Ε, είναι το ίδιο και με τους ξένους μαχητές. Κάθε φιλανθρωπική οργάνωση είναι υπό στενή παρακολούθηση και ξέρουμε ότι το Ισλάμ στην φωσνία Ριζεγοφίνη δεν ήταν ποτέ το βίο Ισλάμ. Ήταν το μετριοπαθές Ισλάμ όπως το λέμε. Τα περισσότερα προβλήματα που είχαμε ήταν εισαγόμενα. Γι' αυτό συνεχίζουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση. Είναι πολύ σημαντικό να σας πω ότι για τους ξένους μαχητές η Βοσνία Ριζεγοβίνη ήταν μία από τις πρώτες χώρες που εισήγαγε νόμο με κυρώσεις για την ε, στρατολόγηση, την ενεργό συμμετοχή ε, σε αυτές ε, τις δραστηριότητες και την οργάνωσή τους. Νομίζω ότι η απόδειξη είναι το γεγονός ότι το 2016 για πρώτη φορά είχαμε ένα έτος με μηδέν αναχωρήσεις προς άλλες χώρες μαχητών. Για αυτούς που επιστρέφουν, 46 πέρυσι, 26 ήδη έχουν ε, ε, ασκηθεί διώξεις εναντίον τους και οι υπόλοιποι είναι υποστενή παρακολούθηση από τις αστυνομικές αρχές. Επομένως, ε, έχουμε μεγάλη ε, αφοσίωση σε αυτό, επικεντρωνόμαστε και έχουμε παρακολούθηση τις σχέσεις μας με το Ηνωμένο Βασίλειο. Ξέρετε, ο κύριος Τζόνσον ήρθε στο Σαράγεβο πριν από μερικές ημέρες. Πολύ καλή συνάντηση. Μπορώ να σας πω ότι δεν το συζητήσαμε και ούτε εμείς είμαστε αυτοί που θα αποφασίσουμε φυσικά το 2018 για την ε, διάσκεψη των δωρητών, όμως εμείς ε, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να γίνει στο Λονδίνο. Ξέρω ότι υπάρχουν κάποιες ιδέες, κάποια διλήμματα. Ο κόσμος λέει εντάξει, τι μήνυμα όμως στέλνουμε. Το Λονδίνο βγαίνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εμείς μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ελοκλήρωση στο Λονδίνο. Η αλήθεια είναι ότι όλες οι χώρες της περιφέρειας και κυρίως η Βοσνία ερσεγοβινη ενδιαφέρονται για τη συνέχιση και την εμβάθυνση των σχέσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο, ακόμα και αν αυτή τη στιγμή είναι στη διαδικασία απένταξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πάνε σε άλλο πλανήτη, σε άλλο κομμάτι της γης, εκεί παραμένουν. Θέλουμε να συνεχίσουμε λοιπόν τις σχέσεις μας. Αν με ρωτάτε λοιπόν για τις σχέσεις μας, αυτό θέλουμε να έχουμε με το Ηνωμένο Βασίλειο. Για το ποιος θα ε, φιλοξενήσει τη διάσκεψη του 2018 δεν μπορώ εγώ να σας δώσω την έγκρισή μου, αλλά για μας δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και είμαστε ευγνώμονε στη Γερμανία και στο Ηνωμένο Βασίλειο που ξεκίνησαν αυτή τη νέα σχέση με τη Βοσνία Ριζεγοβίνη η οποία μας οδήγησε πίσω στις μεταρρυθμίσεις, ε, την διαδικασία ολοκλήρωσης και ένταξης. Ξεκίνησε στο Βερολίνο, ελπίζουμε να τελειώσει αυτός ο πενταετής κύκλος στο Λονδίνο και να δούμε τι θα γίνει. Ε, δική σας όμως απόφαση. Τώρα για το μηχανισμό συντονισμού του κυρίου Ράντος ε, απάντησα πριν. Τώρα για τη δική σας ερώτηση για τα τελωνία. Φυσικά είμαστε υπέρ οποιασδήποτε κοινή δράση. Έτσι το βλέπουμε. Στο Συμβούλιο των Υπουργών μας δεν το έχουμε συζητήσει μεν, αλλά ξέρω ποια είναι η ατμόσφαιρα και πώς ε, το βλέπουν το θέμα η βασική πολιτική. Το υποστηρίζουμε λοιπόν. αν ε, δεν πετύχει, δεν θα φταίμε εμείς. Υπάρχουν κάποιες εξελίξεις σε άλλους παίχτες των Δυτικών Βαλκανίων. Οπότε περισσότερο αυτή είναι το θέμα. Εμείς είμαστε θετικοί. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ για όλες αυτές τις απαντήσεις που μας δώσατε. Μπορούμε να περάσουμε σε ένα δεύτερο γύρο ερωτήσεων. Θα ήθελα στις 11 να έχουμε ολοκληρώσει, γιατί μετέχουμε τον κύριο Ίνσκο. Έχω 8 συναδέρφους στον επόμενο γύρο, 1,5 λεπτό το πολύ ο καθένας, παρακαλώ. Ο αντιπρόεδρος ή αντιπρόεδρος Σουίτσα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ουσιαστικά έχετε απαντήσει στην ερώτηση που ήθελα να θέσω. Έχω κάπως διαφορετικά δεδομένα εγώ για τους ξένους μαχητές, αλλά εσείς έχετε διαφορετικά δεδομένα από τα δικά μου. Τόσο το καλύτερο που είπατε, μηδέν έχουν φύγει από τη Βοσνία σήμερα. Τώρα, μετά το είπε ο κύριος Μακάλιστερ, εγώ είμαι κατά μια ένωσης μέσα στην Ένωση, ότι δεν είναι ο σωστός δρόμος. Θέλουμε η Βοσνία Ζεγοβίνη και όλες οι άλλες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων να ενταχθούν βάσει των κανόνων που ισχύουν. Και έτσι καλώς είναι ο εκλογικός νόμος της Βοσνίας Ερζεγοβίνης που αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου όλοι οι λαοί που συνθέτουν τη χώρα επίσης όρις να μπορέσουν να συμμετέχουν. Δεν αμφιβάλλω για τις επιτυχίες σας. Είπατε ότι υπάρχουν ε, διαφορές που είχαμε στο παρελθόν, αλλά τώρα πρέπει να στραφούμε προς το μέλλον. Πράγματι, αν όμως δεν καταφέρνουμε να τα βγάλουμε πέρα ούτε καν με τον κανονισμό που διέπει τον τρόπο λειτουργίας και τις σχέσεις της Βοσνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, θα έπρεπε να υποφεληθείτε από την ευκαιρία αυτή που έχετε τη στήριξη της Κροατίας και όλων των παραγόντων ε, και ημών των ιδίων εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου να τα καταφέρετε. Πρέπει να συνεργαστούμε για να λυθεί αυτό το ζήτημα. Η ερώτηση πάντως τώρα που θέλω να υποβάλω, μάλλον που ήθελα να υποβάλω, σας είπα ότι απαντήθηκε, οπότε δεν έχω άλλη ερώτηση. Είναι καλό να είναι κανείς αισιόδοξο, αλλά πρέπει μέσα στη Βοσνία Ζεγοβίνη να φροντίσετε για το διάλογο. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Φρόιντ έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ. Εκ μέρου τη Τζούλι Βόρτ, η οποία ζητά συγγνώμη που δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα, ενώ είναι στην αντιπροσωπεία για τη σχέση Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Θέλω όμως να ενισχύσω τις σχέσεις μου με το λαό και την χώρα. Ο λόγος για τον οποίο δεν είμαι εδώ σήμερα είναι ότι είμαι στην Ιταλία με κάποιους νέους από τους πιο λαμπρούς νέους της Βοσνίας Ζεγοβίνης για την πρόθεση της δημοκρατίας μέσω της τέχνης της δημιουργικότητας. Τέτοια προγράμματα δείχνουν πόσα καλά μπορεί να τα καταφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση τι θα ήθελα να πω σε αυτήν την ε, συνάντηση. Αυτό ακριβώς, αυτό είναι το μήνυμά μου. Και ευχαριστώ τον Υπουργό που είναι ανοιχτό, άκουσε το μήνυμα μου αυτό. Ευχαριστώ πολύ, λέει και τον κύριο Ίντσκο που θα έρθει σε λίγο. Είναι καλό να υποφεληθούμε από τις ευκαιρίες που προσφέρονται προς την νεολαία της χώρας. Σας ζητώ να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στους νέους. Ξέρουν τι θέλουν, έχουν τις δυνατότητες, τη γνώση, το ταλέντο και έχουν και προγράμματα. Δεν δραστηριοποιείται βέβαια κάθε νέος, αλλά υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι της νεολαίας που φαίνεται να θέλει να κινητοποιηθεί. Οι νέοι είναι το μέλλον. Δεν πρέπει να τους ξεχάσετε, να μην χάσουν ελπίδα. Είναι ό,τι καλύτερο για όλους αν μας στηρίξετε και στηρίξετε τους νέους στο ταξίδι αυτό. Σάντρα, Τζάρε, Μάριο, Μίλιτσα, Ειρήνα, Ισμύρ και Μιλένα είναι οι νέοι που συνοδεύουν την συνάδελφο στην Ιταλία. Ευχαριστούμε κύριε Φρόντο. Κύριος Βάγκλ τώρα από τους φιλελεύθερους. Ευχαριστώ πρόεδρε και εγώ Υπουργέ, σας καλωσορίζω στην συνάντησή μας και φυσικά και ευχόμαι ότι καλύτερο στο λαό της Βοσνίας Ερζεγοβίνης και στη χώρα σας τα θέματα των συνόρων και των ε, σχέσεων μεταξύ των διαφόρων εθνοτήτων είναι ζητήματα που απασχολούν βέβαια τα Δυτικά Βαλκάνια και ε, δυστυχώς έχουμε λόγους να ανησυχούμε για την τρέχουσα κατάσταση και στα Δυτικά Βαλκάνια και όχι μόνο στη Βοσνία Ερζεγοβίνη, γενικά στα Δυτικά Βαλκάνια. Οι ερωτήσει μου είναι εξή. Πόσο μακριά έχετε καταφέρει να πάτε στι συνομιλίε σα όσον αφορά την οριοθέτηση οριστικά των ε, συνόρων με τις γείτονες χώρες. Και πιο συγκεκριμένα, συμφωνείτε με τους Κροάτες τελικά για την κατάσταση στη γέφυρα, την Νέου. Εγώ θέλω να ξαναπάσω τον Πρόβνικ και ελπίζω να υπάρχει λύση από αυτού όσο γίνεται πιο γρήγορα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Βάγκα. Ο κύριος Κουκάν. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Χαίρομαι που σας βλέπω κύριε Υπουργέ, έρχεται συχνά, οπότε χαιρόμαστε που έχουμε ένα τόσο καλό διάλογο ανάμεσα σε εσά, την αντιπροσωπή για τη σχέση με τη χώρα σα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και γενικά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε ότι μπορείτε να στηρίζεστε σε εμά. Πριν από μερικέ εβδομάδε εγκρίναμε ένα ψήφισμα για τη Βοσνία Ζεγοβίνη, το οποίο καταγράφει κάποια θετικά και συγκεκριμένα βήματα που έχουν γίνει και που δείχνουν ότι η πρόοδος υπάρχει και άρα μπορείτε να προχωρήσετε. Είναι ζωτική σημασία για τις μελλοντικέ εξελίξεις να προχωρήσετε σε αυτό το δρόμο. Τώρα, 77% έχει το κεκτημένο της ΚΠΑ η Βοσνία Ερζεγοβίνη και ελπίζουμε ότι θα μπορέσετε να συνεχίσετε προς αυτή την κατεύθυνση. Ξέρω ότι για να αλλάξει η κατάσταση και η του κόσμου στη Βοσνία Ερζεγοβίνη χρειάζεται χρόνος, αλλά πιστεύω ότι έχουμε περιμένει ήδη πάρα πολύ καιρό και πρέπει να βελτιωθεί η τύχη των ανθρώπων εκεί. Τα είπαν και συνάδελφοι. Εγώ το λέω ότι είναι ο κύκλος της αδράνειας μεταξύ εκλογών. Όταν υπάρχει προεκλογική εκστρατεία, όλα δουλεύουν σε πάρα πολύ χαμηλούς ρυθμούς και δεν υπάρχουν εξελίξεις. Και επειδή υπάρχουν πολλές εκλογές στη Βοσνία Ερζεγοβίνη, αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Μπορεί να γίνει κάτι, ξέρω ότι είναι δύσκολο. Ευχαριστούμε, Έντουερτ. Κύριε Ζόφκο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, παίρνω το λόγο μετά από τον κύριο Κούκαν, ο οποίος ε, βασικά μου πήρε τις λέξεις από το στόμα, γιατί ακριβώς αυτή ήταν και η δικιά μου ερώτηση. Όσον αφορά την απόφαση του Σταγματικού Δικαστηρίου της Βοσνίας Ερζεγοβίνης την Περσινή για την αλλαγή του εκλογικού νόμου Όσον αφορά λοιπόν τον εκλογικό νόμο και τις τροποποίησεις που πρέπει να γίνουν για καλύτερη αντιπροσωπευτικότητα, θέλω να σας ρωτήσω κατά πόσο η απόφαση αυτή θα εφαρμοστεί γρήγορα και αν γίνονται οι προσπάθειες που πρέπει προς αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχει και το πρόσφατο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αναφέρει ε, προβλήματα που έχουν να κάνουν με την απόφαση του στεγματικού Δικαστηρίου, δηλαδή την αλλαγή του εκλογικού νόμου, τις αλλαγές στη πόλη του Μόσταρ και που ζητάει και μεταξύ άλλων και πιο μεγαλύτερο πλουραλισμό των μέσων ενημέρωση. Μπορείτε λοιπόν να μας πείτε πού βρισκόμαστε σε σχέση με τη λύση των προβλημάτων αυτών. Και θέλω να ρωτήσω και την είπα το εκπρόσωπο. Τι σκοπεύει να κάνει για να προχωρήσουμε προς τη λύση αυτών των δυσκολιών. Πρόεδρος. Ωραία. Πίτια. Προχωράμε στους τρεις τελευταίους ομιλητές μας δηλαδή. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, Η πρόοδος που καταγράφει η Βοσνία Ερζεγοβίνη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πράγματα που βρίσκω θετικά και με χαροποιούν. Χρειάζονται και άλλες προσπάθειες αν θέλουμε να υλοποιηθούν πλήρως οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Αναφέρθηκε το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε πρόσφατα. Εκεί μιλάμε για την τροποποίηση του εκλογικού νόμου και για τη δυνατότητα ενός ομοσπονδιακού μοντέλου που θα χειρίστε με τον ίδιο τρόπο όλες τις ε, εθνότητες. Υπάρχει και το θέμα όμως της προστασίας του περιβάλλοντος και υπάρχει απόφαση και από αυτού. Υπάρχει πρόοδος λοιπόν στη χώρα όσον αφορά την βελτίωση της λειτουργίας του δηληστηρίου που από όσο ξέρουμε έχει καταστροφικές συνέπειες η λειτουργία του σταθμού αυτού στον κόσμο και στους Κροάτες μάλιστα που ζουν στην Κροατία. Ευχαριστούμε κύριο Νάρτ από τους φιλελεύθερου. Ευχαριστώ πρόεδρε. Στη Βοσνία Αρζεγοβίνα έχουμε το θέατρο, δηλαδή όλη αυτή την υπερδομή, τις φιλοσοφικές, ρητορικές, όλα αυτά που προχωρούν, νομιμότητα, ναι, αλλά υπάρχει και η πραγματικότητα και αυτό το λέμε πολύ πόνο. Η Βοσνία Αρζεγοβίνη γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι δεν υπάρχει. Υπάρχουν τρει κοινότητε, οι οποίε ήταν σε πόλεμο μεταξύ του και τώρα έχουν γυρίσει η μία την πλάτη στην άλλη. Δεν υπάρχει σχέση μεταξύ των διαφόρων συστατικών τη Βοσνίας Αρζεγοβίνη. Οπότε έχουμε να κάνουμε με ένα τεχνητό κράτο που επιπλέον έχει εσωτερικά προβλήματα που στηρίζονται και από εξωτερικούς παράγοντε Ούτε η Κροατία ούτε η Σερβία βοηθούν την κατάσταση. Κάθε άλλο. Ούτε και η Μακεδονία, ας πούμε, βοηθάει την Βολγαρία ή την Αλβανία ή την Ελλάδα. Συνεπώς, έχουμε να κάνουμε με μια κατάσταση όπου η πολιτική μεταφυσική που μπορεί να είναι οι δηλώσεις μας, οι διατυπώσεις εξαιρετικών νόμων, τελικά δεν εξυπηρώνουν απολύτω τίποτα. Γιατί η πραγματικότητα είναι ότι οι κοινότητε αυτέ εξακολουθούν να έχουν γυρισμένη την πλάτη μεν στου δε. Δεν υπάρχει χώρα. Και το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και για μένα πάρα πολύ ευαίσθητο γιατί υπάρχει κίνδυνος έκρηξης όπως υπάρχει στη Μακεδονία. Λέει ο στη η Μακεδονία είναι πιο έντονο. Οπότε ρωτάω πόσοι νόμοι χρειάζονται ακόμα, πόσοι κανονισμοί, πόσα υπουργεία ακόμα θα δημιουργηθούν μέσα σε αυτή την έκρηξη από τον πολυάριθμο, τα πολυάριθμα υπουργεία προκειμένου κοινωνικά τελικά να υπάρξει αυτή η χώρα, η Βοσνία Ερζεγοβίνη. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Πέτερλε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τα, καλά, για τα λόγια σας και για την ευρωπαϊκή φιλοδοξία που πάντα είναι ευπρόσδεκτη εδώ. Νομίζω πως η χώρα σας πρώτα απ' όλα έχει να αντιμετωπίσει την εξή πρόκληση. Πώ θα μπορέσει να σταθεί ενωμένη μέσα στην διαφορετικότητα. Και εσείς είπατε κάτι πολύ σημαντικό. Η ειρήνη δεν είναι η απουσία πολέμου. Η απουσία πολέμου είναι σημαντική, αλλά όχι η επαρκής. Και τη δεύτερη παρατήρηση εσείς ήταν η συνεργασία. Η μελλοντική ευρωπαϊκή προοπτική της Βοσνίας Ριζεγοβίνης και ολόκληρης της περιοχής εξαρτάται από αυτήν την συνεργασία. Και το ερώτημά μου είναι, πού πιστεύετε ότι μπορούμε να περιμένουμε πιο δυναμική προσέγγιση ως προς αυτήν την κατεύθυνση στη χώρα και πώς βλέπετε την ιδέα μιας νέας αγοράς των Δυτικών Βαλκανίων Κάποιοι λένε ότι θα ήταν δυνατόν ε, να επιτευχθεί μέσα σε τρία χρόνια κάτι τέτοιο. Και έπειτα το σχόλιο μου για το τον Τζόνσον και το Λονδίνο. Εγώ συμφωνώ μαζί σας. Δεν περιόριζα το Ηνωμένο Βασίλειο που είναι ακόμα μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης με όλα τα δικαιώματα και τα καθήκοντα ε, όσον αφορά την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, έχετε τώρα έξι λεπτά για να απαντήσετε αυτό το δεύτερο γύρο. Καλή τύχη. Μάλλον καλή επιτυχία. Ε, ναι, δεν ξέρω κατά πόσο είναι δυνατό κάτι τέτοιο, αλλά θα προσπαθήσω. Καταρχά ε, για την κυρία Σουίτσα, το θέμα για τους μηδέν ξένου μαχητές που φεύγουν από τη Βοσνία για ξένα πεδία μάχης, αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία που έχουμε από το Υπουργείο Ασφαλεία τη χώρα μου. Το θέμα της ενίας αγοράς και των ε, τελωνίων εδώ έγιναν διάφορα σχόλια. Βεβαίως δεν μπήκα στις λεπτομέρειες, αλλά εμείς αυτό το αντιλαμβανόμαστε ως κάτι που μας βοηθά να συνεχίσουμε την ευρωπαϊκή μας πορεία είναι ένα υποκατάστατο για την ένταξή μας, όχι μόνο για την Βοσνία Ριζαγοβίνη, αλλά όλες οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων θα ήταν κατά. Δεν μπορεί αυτό να υποκαταστήσει την ένταξη. Μπορεί να είναι ένα εργαλείο για να κινηθούμε πιο γρήγορα. Ο εκλογικός νόμος. Ναι, βεβαίως. Καλό όλους τους, ε, τους ε, φορείς να βρουν λύση, γιατί δεν είναι τώρα αν θέλουμε ή δεν θέλουμε να το κάνουμε, είναι και ο κανόνας του συνταγματικού δικαστηρίου. Αλλά και πάλι πρέπει να γνωρίζουμε. Και γι' αυτό θα είμαι πολύ άμεσος και έντιμος ότι αυτό εξαρτάται από τους παίχτες στην Ομοσπονδία της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, δηλαδή την Ομοσπονδία μεταξύ Βοσνίων και Κροατών γιατί πρέπει να δούμε πώς θα βρεθεί ο τρόπος ώστε οι διεφθαρμένοι Μάλλον, συγγνώμη, ώστε οι, ε, οι λαοί να μπορούν να εκλέξουν τους εκπροσώπους τους. Ε, όχι μόνο στο Εθνικό Κοινοβούλιο, αλλά και ε, στα περιφερειακά. Συμφωνώ ότι χρειάζεται περισσότερη δράση από την κυβέρνηση και από τις διάφορες δομές ε, της χώρας ε, αλλά και περισσότερη δράση ναι, από τους νέους. Να ξυπνήσει το επιχειρηματικό πνεύμα των νέων. Μία από τις πρόσφατες έρευνες έδειξε ότι το 97% των νέων στα, στα σχολεία τι θέλουν να κάνουν, να δουλέψουν για την κυβέρνηση, για την πόλη, για το Δήμο ή για τους φορείς τηλεπικοινωνιών. Δεν σκέφτονται για τίποτα δικό τους, για δικά τους project. Για τα σύνορα, ναι. Τελειώσαμε με το Μαυροβούνιο. Πριν από 1,5 χρόνο το υπογράψαμε. Συζητάμε με την Κροατία και την ε, Σερβία. Δεν έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα που να δημιουργηθούν προβλήματα ασφάλειας ανάμεσα στις χώρες. Συνεχίζονται οι διαδικασίες λοιπόν. Τώρα για τη γέφυρα Πέρεζα έχουμε βρει λύση. Εξ αρχής πίστευα ότι, ότι ήταν τεχνικό θέμα. Και τώρα ε, ξέρουμε πως ήταν θέμα της προηγούμενης ε, κυβέρνησης ε, της Κροατίας και τότε μετετράπησε σε πολιτικό ζήτημα και αν επανέλθουμε στην τεχνική φύση του ζητήματος θα βρούμε λύση. Γιατί είναι δύο φιλικές χώρες που συναντώνται στην γέφυρα ο καθένας με τα συμφέροντά του. Η Κροατία βεβαίως, που είναι φυσιολογικό, θέλει να συνδέσει κομμάτια της δικής της επικράτειας. Η Βοσνία Ζεγοβίνη επίσης, πράγμα που είναι φυσιολογικό, θέλει να προχωρήσει προς την ανοιχτή θάλασσα. Η ιδέα είναι λοιπόν πώς θα βρούμε κοινό έδαφος ώστε να ανταποκριθούμε σε όλα τα συμφέροντα. Έτσι κι αλλιώς η γέφυρα δεν θα χτιστεί και τόσο σύντομα. Ελάτε λοιπόν και φέτος Ευχαριστώ τον κύριο Κούκαν για τα σχόλιά του για τη Βοσνία και τον λαό μας. Ναι, έχουμε πολλές εκλογές. Τι μπορούμε να κάνουμε και αυτή είναι μια ιδέα για την αλλαγή του εκλογικού νόμου, δηλαδή να έχουμε τις τοπικές και τις γενικές μαζί. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε. Θα είναι περίπλοκο, αλλά μπορεί να γίνει. Ε, να έχουμε έτσι δηλαδή μία ταυτόχρονη τετραετία. Επίσης ρωτήσατε για το ψήφισμα και τι θα κάνουμε για τα θέματα του Μοστάκ της ελευθερίας του τύπου και ένα κανάλι με την κροτική γλώσσα. Όλα αυτά είναι κρεμή. Χρόνια τώρα είναι αυτά τα θέματα μας απασχολούν. Υπάρχουν μηχανισμοί για να τα αντιμετωπίσουμε, αλλά χρειάζονται λύσεις, λύσεις εσωτερικές. Μια εσωτερική συμφωνία είναι, νομίζω, απαραίτητη. Κυρία Πετήρ, ναι, οικολογία πολύ σημαντικό θέμα για μας. ιδιαίτερα αυτό της ρήπανσης ε, στις πόλεις. Ε, στο συνεζήτησαμε και με τον Υπουργό της Κροατίας. Μετά είχα συνομιλίες με ε, ανώτατους αξιωματούχους της κυβέρνησης της Σερβίας, με τον Υπουργό Μπόριτς και εκείνη είναι υπέρ της συνεργασίας. μία λύση είναι ο περιορισμός του δηληστηρίου. Δεν λέω για άλλα κομμάτια στη Βοσνία, αλλά εν πάση περιπτώσει να αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας του δηληστηρίου ώστε να μειωθεί η ρήπανση. Τουλάχιστον για αυτή τη φάση, από ό,τι εγώ κατάλαβα, αυτό θα γίνει με το, στη συζητήση με τον κύριο Στυρ. Αυτό θα είναι ικανοποιητικό για τον κόσμο του ρόλου, γιατί όλοι υποφέρουν από αυτό. Κύριε Νάρτα μου, είχαμε πολύ... Μιλήσατε με πολύ έντονα λόγια, αλλά αισθάνθηκα ότι με καλή την πρόθεση τα είπατε όλα αυτά και το, το μήνυμα κλειδί είναι κάτι που θέλω και εγώ να επαναλάβω. Εδώ πρέπει να είμαστε περισσότερο στραμμένοι προς, ο ένας προς τον άλλον, όχι με την πλάτη ο ένας τον άλλον. Δηλαδή τρεις κοινότητες να είμαστε ένα να μιλήσουμε περισσότερο μεταξύ μας και σίγουρα εγώ ε, συμμερίζομαι την ανησυχία σας για την ε, Μακεδονία. Ε, το μόνο που πρέπει να πω ότι διαφωνώ, αν κατάλαβα καλά βέβαια τα σχολιά σας, είναι ο ρόλος του Βελιγραδίου για του Ζάγκρεπ. Δεν νομίζω ότι είναι κομμάτι του προβλήματος. Η ανησυχία των Κροατών και των Σέρβων είναι φυσιολογική. Και η προσέγγιση αυτή είναι επικοδομητική. Είχαμε μια κοινή συνεδρίαση και με την κυβέρνηση της Σερβίας. Θα γίνει και κοινή συνεδρίαση αρχές Ιουνίου με την κυβέρνηση της Κροατίας και σύντομα θα μπορέσουμε να εστιάσουμε σε θέματα πραγματικά. Τέλος, ο κύριος Πέτερλε με ρώτησε πότε θα συνεργαστούν περισσότερο. Ε, αυτό, είναι, αυτό είναι το θέμα για τη χώρα μου. Ότι, δηλαδή, ακόμα ελπίζω πως και αυτές οι ε, ε, ε, συνομιλίες για τον εκλογικό νόμο και την ατζέντα των μεταρρυθμίσεων θα μας δώσει θετική απάντηση για όλα αυτά. Βεβαίως, έχω ήδη μιλήσει για αυτή την ιδέα της κοινή αγοράς, των τελωνίων κτλ. Επαναλαμβάνω ότι είναι σημαντικό για μας εάν συμβεί κάτι τέτοιο. Εμείς το βλέπουμε ως μια βοήθεια για να επιτεχυνθεί η διαδικασία, όχι ως υποκατάστατο για την ένταξη της χώρας μας στην Ένωση. Κύριε Τσέρνακ, ε, να, κάνω, να σας ευχαριστήσω καταρχάς που ήρθατε για αυτή την ανταλλαγή απόψεων που απαντήσατε στις ερωτήσεις μας και μας δώσατε πολύτιμες πληροφορίες. Δεύτερον, να ζητήσω συγγνώμη που δεν γράψαμε σωστά το όνομά σας εκεί. Ξεχάσαμε ένα α. Είναι Τσέρνεντακ. Τσέρνεντακ και όχι Τσέρνεντακ, που είναι γραμμένο λάθος. Και να σας ευχαριστήσω λοιπόν εξ ονόματος ολόκληρης της Επιτροπής. Θα διατηρήσουμε τον επικοδομητικό διάλογο μαζί σας και με άλλους ε, προσώπους της χώρας σας. Να επιβεβαιώσω επίσης ε, Υπουργέ και κυρία Πρέσβη ότι η Επιτροπή μας θα συνεχίσει να στηρίζει την Βοσνία Ερζεγοβίνη ε, όπως το αξίζει. Σας ευχαριστώ που ήρθατε και εύχομαι να περάσετε καλά στις Βρυξέλλες. Ωραία λοιπόν κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ. Γεια σας ε, Υπουργέ, γεια σας ε, κυρία Πρέσβη. Θα τα ξαναπούμε σύντομα και τώρα περνάμε στο επόμενο μας θέμα που είναι και πάλι Βοσνία Ριζεγοβίνη και θα ήθελα τώρα να ζητήσω από τον ε, κύριο Βαλεντινέσκο να έρθει εδώ. Από τον κύριο Βαλεντίν Ίσκο να έρθει εδώ στο έδρανο του Προεδρείου. Herzlich willkommen. Chris Gott, danke für den schönen Empfang. Ja, wo sitze ich? Sie sitzen hier. So. Lieber Ensko, herzlich willkommen. Ladies and gentlemen. Κύριε Ιβανιέσκου, καλώ ήλθατε. Κυρίε και κύριοι, πάμε στο σημείο 14 τη ημερήσια διάταξη. Καλωσορίζω τον κύριο Βαλεντίν Ινσκού που είναι ο ύπατος εκπρόσωπος του ΟΗΕ για τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Ας πούμε ότι είναι ο θεματοφύλακας ε, της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Ακούσατε ήδη τη συζήτηση με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Τσέρνεντακ. Είδατε ποιες είναι οι ερωτήσεις που έθεσαν οι συνάδελφοι. Άρα, χωρίς άλλη καθυστέρηση, να δώσω σε εσά το λόγο για 10 λεπτά περίπου και μετά για άλλη μια φορά θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τα σημεία που μας ενδιαφέρουν. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι και τόσο εύκολο να μιλήσει κανείς ε, σε 10 λεπτά για μια χώρα που έχει 14 κυβερνήσεις, ε, τρεις ε, θρησκείες, ε, τέσσερις εθνότητες, ε, πολλές γραφές και μία ελπίζω διεθνή κοινότητα. Υπάρχουν πολλές οι προκλήσεις λοιπόν. Η κατάσταση έχει αλλάξει πολύ από το 1990 και μετά. Οι απειλές όμως για τη σταθερότητα υφίστανται ακόμα. Βασικά αυτές οι απειλές βρίσκονται στη διχαστική πολιτική κάποιων πολιτικών κομμάτων, στην κλεπτοκρατία και φυσικά αυτές οι πολιτικές δεν βοηθούν το μέλλον της Βοσνίας Αρζεγοβίνης οι ηγέτες κάποιων πολιτικών κομμάτων απλώς διατηρούν τα προνόμια τους. Αναγνωρίζουμε λοιπόν αυτά το οικονομικό κίνητρο για τους περισσότερους πολιτικούς ως την πηγή του προβλήματος. Όμως τελικά υπάρχει κάτι που απειλεί περισσότερο τη σταθερότητα. Μια συνεχής ρηγμάτωση και κατακαιρματισμός της χώρας σε εθνοτικό επίπεδο η πρόσφατη πρόοδος της Βοσνίας Ερζεγοβίνης στη διαδικασία για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι βέβαια το αντίθετο. Είναι ιδιαίτερα επιτυχημένη από το 2016 και μετά. Αν μιλήσουμε τώρα για το μέλλον της χώρας, θα πω ότι είναι καλό ε, να υπάρχει πρώιμη ε, αποδοχή της υποψηφιότητας και ύστερη ένταξη όταν υπάρξουν ε, οι κατάλληλες συνθήκες και έχουν εκπληρωθεί τα οι όροι. Εγώ συγκεκριμένα είμαι υπέρ ενός σχεδίου δράσης ε, που ε, θα οδηγήσει την Βοσνία Αρσεγοβίνη στην αίθουσα απομνήσει και για τον ΝΑΤΟ. Οι απόψει μου για την Βοσνία ε, υφίστανται λόγω της εμπειρίας μου τα τελευταία 8 χρόνια ως είπατε ως εκπρόσωπος. Βλέποτε στάσεις γενικά όλο αυτό το διάστημα, όχι τα τελευταία, το τελευταίο διάστημα. Η διχαστική και αποσχεστική ρητορική έχει γίνει ε, πολύ ουσιαστική και υπάρχουν ε, διχαστικά ζητήματα όπως ε, είναι η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για κάποιους πολιτικούς ε, πριν από 25 χρόνια είχαμε ακριβώς την ίδια στάση που οδήγησε στον πόλεμο. Δυστυχώς ε, το κράτος δικαίου ε, δεν υφίσταται διότι οι πολιτικοί αγνοούν τις δικαστικές αποφάσεις και ασκούν και πίεση στους δικαστές. Τα δικαιώματα των πολιτών ε, είναι κάτι που τη χάνει συνεχώς άρνησης Και ειδικά μετά τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ε, δεν έχει ακόμα δικαιωθεί ο κόσμος που θέλει να έχει κάποιες δημόσιες θέσεις. Επίσης, ε, το Διεθνές Επιδημικό Δικαστήριο ανέδειξε ακριβώς πώς η Προεδρία και όλοι οι θεσμοί μπορούν να αναδειχτούν σε ένα όπλο. Οι πολιτικές δυνάμεις βέβαια ήταν προμηθείς όταν ε, έπρεπε να κάνουν πολιτικές ε, οπισθοδρομικές. Δεν δίνουν δικαιώματα σε μικρότερες εθνοτικές ομάδες και γλωσσικές ομάδες για να ε, είναι στο σχολείο, ας πούμε, στο Άιτσε, σε μια κεντρική πόλη της Βοσνίας. Είχαμε διαμαρτυρίες ε, μαθητών που διαμαρτύρονταν κατά του διαχωρισμού των μαθητών στο σχολείο μετά από πολλά χρόνια έγινε κάτι τέτοιο και πάλι. Αυτό δεν είναι καλό για το μέλλον της χώρας, όχι όμως ε, για τους πολιτικούς ε, και τους δικούς τους οι άνθρωποι, ο λαός έχουν μεγάλη ανησυχία και όσοι πλήττονται φεύγουν από τη χώρα, ενώ οι ξένες επενδύσεις μειώνονται. Όλα αυτά είναι σε αντίθεση με τα όσα ε, ε, ίσχυαν το 2006 που η χώρα ήταν γεμάτη εμπιστοσύνη στον εαυτό της και ενθουσιασμό. Είχαμε τρεις στρατούς ε, πριν από 11 χρόνια. Τώρα έχουμε ένα Υπουργείο Άμυνας, μια υπηρεσία πληροφοριών, μια σημαία που δεν είχαμε, ένα καλό και ισχυρό νόμισμα, συνοριοφυλακή κτλ. Η διεθνής λοιπόν κοινότητα ήταν πολύ επιτυχημένη τα πρώτα δέκα χρόνια. Ήταν έτοιμη να προωθήσει φιλόδοξες πολιτικές που οι πολιτικοί της χώρας πίστηκαν ότι άξιζαν τον κόπο. Το συμπέρασμά μου σήμερα βέβαια είναι ότι η διεθνής ε, κοινότητα γίνεται όλο και πιο ασθενής και κουρασμένη δεν θα κάτσουν εκεί να περιμένουν, θα, ε, γιατί η στάση των πολιτικών είναι ότι απλώς θα βαρεθούν να μας ε, αντέχουν. Φαίνεται λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ενισχύσει τις ε, δραστηριότητες της και να δώσουμε ένα αίσθημα επίγοντος στη χώρα. Χρειάζεται μια στρατηγική επανεμπλοκή έτσι ώστε να αλλάξουν τα πράγματα στη Βοσνία ριζεγοβιν Καταρχάς, ε, η χώρα αυτή είναι μια χώρα η οποία είναι δυνατόν να ευημερήσει και είναι πολύ σημαντική για τη σταθερότητα της Ευρώπης. Ο πρόεδρος Βούτσιτς που πρόσφατα εξελέγει το ε, καταλαβαίνει αυτό και γι' αυτό οδήγησε και τη Σερβία προς την Ευρώπη. Ο, ο Πρωθυπουργός Πλάνκοβιτς ε, της Κροατίας επίσης είναι υπέρμαχος της σταθερότητας στην περιοχή και έχει βοηθήσει, έχει προσφέρει χειραβοήθειας ε, στην Βοσνία Ερζεγοβίνη πολλές φορές στο παρελθόν. Η χώρα επίσης όπως και η Ευρώπη είναι μια πολυεθνική ε, κοινωνία με πολλές ε, θρησκείες. Έχουμε εδώ και 400 χρόνια τόσες πολλές θρησκείες, όμως ο κόσμος έχει μάθει να ζει, να συμβιώνει. Υπάρχει ανοχή και υπάρχει ευρωπαϊκός τρόπος ζωής στην Βοσνία Ερσεγοβίνη. Τρίτον, πρέπει να δούμε εμείς ε, τα λάθη μας ως Ευρωπαϊκή Ένωση στο παρελθόν που συνεισέφεραν στα τραγικά γεγονότα στη Βοσνία Ερσεγοφίνη. Έχουμε ηθικό καθήκον να ακολουθούμε τις αξίες μας για να πετύχουμε το επιθυμητό. Η Βοσνία Ερσεγοβίνη θέλει να στείλει ένα μήνυμα στις άλλες χώρες ότι έχει κάνει τη σωστή επιλογή ε, στις στρατηγικές της προτεραιότητες ζητώντας να μπει στην οικογένεια της Ευρωπαϊκής. Τώρα που γιορτάζουμε την 60η επέτειο της συνθήκης της ε, Ρώμης, θα θυμηθείτε που ήσασταν εσείς μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τι ακριβώς είναι η Ευρώπη, η ειρήνη, σταθερότητα και ευημερία μέσα από την Ένωση, όχι την, το διχασμό. Να τονίσω βέβαια ότι υπάρχει ανταγωνισμός. Πρέπει να σταματήσουμε να θεωρούμε ότι ε, επειδή είμαστε, έχουμε δίκιο, επειδή έχουμε δίκιο, δηλαδή όλα θα γίνουν όπως τα λέμε εμείς, φαίνεται σύμφωνα με τον ε, βοσνιακό ε, τύπο ότι η, η, Βοσνία έχει κάνει συμμαχία με τη Ρωσία και έγιναν κάποιες ασκήσεις στο Καζακστάν τον Σεπτέμβριο. Βέβαια, ε, έχουμε ακούσει και τον πρέσβη να λέει ότι η Ρωσία είναι εναλλακτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις ε, με μεγάλη... Ε, ε, με μεγάλη αιμονή για να μπορέσουμε να κάνουμε τη Βοσνία Ερζεγοβίνη ένα λειτουργικό και κράτος, όχι με κεντρική εξουσία απαραίτητα, αλλά να λειτουργεί και να έχει ευημερία. Έχουμε ήδη πετύχει απίστευτες επιτυχίες στη Βοσνία Ερσεγοβίνη επειδή είμαστε αναφοσιωμένοι και φιλόδοξοι. Αν συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό θα επιτύχουμε εκπληκτικά αποτελέσματα. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, Mr. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Ίντσκο για τις παρατηρήσεις σας αυτές. Τώρα, έχουμε 15 λεπτά γιατί βλέπετε σε 10.30 αρχίζει η κοινή ε, συνάντηση που έχουμε με την Επιτροπή Ανάπτυξης και Επιτροπή Προϋπολογισμών. Έχουμε 8 μιλητέ 1,5 λεπτό το πολύ ο καθένας και αρχίζουμε τον κύριο Κούκαν. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε κύριε Ίνσκο. Χαιρόμαστε που σας έχουμε μαζί μας. Υπάρχουν ε, πραγματικά πολύ λίγοι άνθρωποι που έχουν τέτοια θεσμική μνήμη όπως έχετε εσείς για την Βοσνία Ριζεγοβίνη. Σας ευχαριστούμε πολύ λοιπόν που οδηγείτε προς την Ευρώπη τη χώρα και που στηρίζετε την ευτική διαδικασία. Αξίζεται την πλήρη εκτίμησή μας και τον απόλυτο σεβασμό μας. Δύο ερωτήσεις έχω. Μπορείτε να μας πείτε παρακαλώ για την περιφερειακή δυναμική και τις διμερείς σχέσεις της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Έπειτα ποιοι εξωτερικοί παράγοντες πιστεύετε ότι μπορούν να βοηθήσουν ή μπορούν να επηρεάσουν περισσότερο τη χώρα. Και δεύτερον, μπορείτε να σχολιάσετε για τα αποτελέσματα του 2013, την απογραφή που έγινε τότε. Υπάρχει περίπτωση να έχουμε κοινά ε, στοιχεία απογραφής μεταξύ των δύο πλευρών της Ομοσπονδίας δηλαδή και της Ρεπούμπλικας Φρεσκά. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Πίτσουλα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Νίσκο, πάντα σας υποδεχόμαστε με ιδιαίτερη χαρά εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ανταλλάσσουμε μαζί σας απόψεις. Χαίρομαι λοιπόν που είπατε ότι η Βοσνία Ερζεγοβίνη πρέπει να είναι μια χώρα η οποία να λειτουργεί, όχι να είναι κεντρικά δικούμενη. Ποια είναι η πραγματικότητα όμως σήμερα της Βοσνίας Ζεκοβίνη. Dayton, Ευρωπαϊκή Ένωση επηρεάζουν την πορεία της χώρας, οπότε θέλω να ξέρω πόσο ισχυρή, πόσα δύναμη είναι οι θεσμοί στη Βοσνία Θεσμοί οι οποίοι πρέπει να αντικαταστήσουν, έπρεπε να αντικαταστήσουν μάλλον μετά τον πόλεμο της, ε, τη διεθνή βοήθεια και τη δίκηση που υπήρχε εκεί. Ποια είναι η προτεραιότητα, η πρόληψη, η ανάκαμψη ή πραγματικά η διαδικασία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντάξει, μπορούν ίσως να πάνε και παράλληλα όλα αυτά. Αν όχι όμως, και υπάρχουν πολλά που δείχνουν ότι ακόμα υπάρχει μεγάλη πόλωση. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Ράντος. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ίνσκο που είναι μαζί μας εδώ σήμερα. Η ερώτησή μου έχει να κάνει με τις αποφάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου στη Βοσνία Ερζεγοβίνη. που λέει σε επίπεδο των δύο οντοτήτων οι αποφάσεις ισχύουν εξίσου. Όμως ε, δεν λειτουργούν, οπότε είναι σαν να λειτουργεί παράνομα η χώρα. Μία απόφαση λέει ότι η πλειοψηφία στην κάθε πλευρά χέρι των αντιπροσώπων της στο κοινοβούλιο για να υποστηρίξουν ακριβώς τα συμφέροντα των λών Ο τρόπος με τον οποίο αυτό ελοπείται σήμερα όμως είναι σε βάρος της πολιτικής βούλησης του κόσμου και κατά του συντάγματος του ίδιου της Βοσνίας Αρζεγοβίνης. Κάποιοι οποίοι είχαν ε, θέσεις ε, παρενέβησαν. Άλλοι αποφάσισαν να μην παρέμβουν. Θέλω να ακούσω πάντως τα δικά σας σχόλια για αυτήν την κατάσταση που είναι αντισυνταγματική στη Βοσνία Ζεγοβίνη σήμερα. Ευχαριστούμε κυρία Σουίτσα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καλώς ήρθατε κύριε Ινσκό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα είμαι σύντομη. Θέλω να ρωτήσω ποια είναι η δικιά σας εκτίμηση όσον αφορά τις αλλαγές στον εκλογικό νόμο. Πιστεύετε ότι θα υλοποιηθεί? Από όσο ξέρω, δεν μπορεί να συμβεί αυτό ένα έτος εκλογών. Άρα μπορεί να γίνει φέτος. Εσείς τι νομίζετε. Και δεύτερον, έχετε καθόλου αξιόπιστες σφιγμομετρήσεις από τον λαό της Βοσνίας Ζεγοβίνης όσον αφορά τη στάση του απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχετε αξιόπιστα στοιχεία. Και θα έλεγα ότι αν δεν αλλάξει η Βοσνία Ζεκοβίνη, θα έπρεπε να αλλάξει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να αλλάξει τα κριτήριά τη, άρα πρέπει να γίνουν αλλαγέ στη Βοσνία Ζεκοβίνη και να υλοποιηθούν οι μεταρρυθμίσει εκεί. Ευχαριστούμε. κύριο Φρόιντ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ντσκο, που ήρθατε σήμερα. Αν σας κατάλαβα καλά, Ζητάτε η Ευρωπαϊκή Ένωση να παίξει πιο ισχυρό ρόλο στη διαδικασία προσχώρησης και να υπάρξει έτσι μια πιο γρήγορη διαδικασία προσχώρησης τη Βοσνίας Ερζεγοβίνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πράγματα που συζητιούνται και για άλλες χώρες, δεν θέλω τώρα να τις κατονομάσω. Είχε γίνει συζήτηση για το κατά πόσο εμείς πήγαμε υπερβολικά πολύ γρήγορα και το ότι ακριβώς δεν περιμέναμε αρκετά προκειμένου να υπάρξει το κράτος δικαίου, να καταπολεμήσει η χώρα αυτή επαρκώς ε, την διαφθορά, ώστε μετά να γίνει η προσχώρηση αυτή. Και το επιχείρημα ήταν, μα άμα μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι χώρες, τότε θα λυθούν από μόνα τους τα προβλήματα αυτά. Οπότε ερωτώ, είναι αυτός ο σωστός δρόμος? Ποιος είναι ο σωστός δρόμος? Δεν πρέπει να περιμένουμε προκειμένου το ευρωπαϊκό και ότι είναι τόσο σημαντικό για μας την Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρξει στη χώρα και μετά να δεχτούμε τη Βοσνία Ερζεγοβίνη ή πιστεύετε ότι είναι προτιμότερο να μπει η Βοσνία και ό,τι προβλήματα εκκρεμούν να προσπαθήσουμε να τα λύσουμε μετά. Ευχαριστούμε κύριε Φρόντ, ο κύριος Βάγκλ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κυρίνσκο, νομίζω ότι θα με καταλάβετε αν μιλήσω στη μητρική μας, οπότε θα υποβάλω την ερώτησή μου στα σλοβενικά. Έχετε επιδείξει πολύ υπομονή. Και ήσασταν και πολύ επικοδομητικός όλα αυτά τα χρόνια που έχετε περάσει στη Βοσνία Ζεγοβίνη. Νομίζω ότι πρέπει όλοι να εκφράσουμε την εκτίμησή μας στο πρόσωπό σας, γιατί ε, εκθέσατε τον εαυτό σας σε καταστάσεις πολύ, που έχουν ένα συμβολισμό πολύ σημαντικό και αυτός ο συμβολισμός στα Δυτικά Βαλκάνια ήταν το πιο ευαίσθητο. Οι διάφορες ε, πέτοι στην Ρεπούμπλικα Σφρέσκα, Σερβενίτσα κτλ. Ο συμβολισμός αυτός λοιπόν, πιο σημαντικός και από τη ρητορική, μας υπενθυμίζει ότι οι διεθνωτικές σχέσεις είναι ένα ζήτημα που παραμένει σε κρεμότητα. Και η ερώτησή μου είναι η εξής. Εσείς που είσαστε, είπα, εκπρόσωπος του ΟΗΕ, πιστεύετε ότι το συμφέρον της Βοσνίας Ερζεγοβίνης και των Δυτικών ε, Βαλκανίων ε, πιστεύετε, μάλλον ότι το ενδιαφέρον αυτό για αυτά τα συμβολικά είναι κάτι το επαρκές. Ευχαριστούμε. Επόμενο μιλήτρια, ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει η κυρία Ζόφκο. Οι προλαλήσαντε ρώτησαν πολλά από αυτά που ήθελα να ρωτήσω και εγώ, δηλαδή για τον εκλογικό νόμο και για την υλοποίηση των αποφάσεων του Συνταγματικού Δικαστηρίου. Υπενθυμίζω ότι το 2003 εφαρμόστηκαν μεταρρυθμίσεις επειδή οι εκπρόσωποι των Κροατών βοήθησαν. Γιατί λες ποιος θα μπορούσε να εφαρμόσει την αμυντική αυτή μεταρρύθμιση και να δημιουργούσε ένα Υπουργείο Άμυνα σε επίπεδο χώρας και υπηρεσία πληροφοριών. Στη συνέχεια, το 2011, δημιουργήθηκε η πλατφόρμα που θελοποιούσε τις αποφάσεις. Δεν πιστεύετε ότι μην έχοντας την αλλαγή στον εκλογικό νόμο και έχοντας το 2018 μια κατάσταση στην Ομοσπονδία της Βοσνίας Ερζεγοβίνης που θα είναι κρυκτική, δεν θα δημιουργήσει περισσότερη αστάθεια. Πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία αν θέλουμε σταθερή την Βοσνία Ερζεγοβίνη. Πρέπει να υπάρχει νόμιμη εκπροσώπηση στην κυβέρνηση. Και ελπίζω εσείς να λάβετε υπόψη σας όλους τους παράγοντες για να μπορέσετε να καταλήξετε σε συμβασμό. Ευχαριστούμε ο κύριος Γκάλερ. Ευχαριστώ στη Βονζία Έχουμε μία σύραξη με λέξεις. Από τη μία έχουμε το δημοψήφισμα και ε, δεν μπορεί κανείς να το εμποδίσει και αν είμαστε, αν έρθει αυτό το δημοψήφισμα δεν θα μπορεί κανείς να το σταματήσει. Ε, θα γίνει το δεύτερο δημοψήφισμα με 99% έγκριση θα, ανα, θα αναγνωριστεί από τη Ρωσία και θα στείλει ε, τους, ε, το στρατό της για να γνωρίσει αυτό το νέο κράτος ε, και εμείς θα είμαστε γελοί. Τώρα έχουμε στρατεύματα σε μικρό βαθμό αλλά είναι σε ετοιμότητα. Αν δεν μπορεί το Σαράγεβο να το εμποδίσει αυτό θα πρέπει εμείς να το κάνουμε. Το θέμα είναι αν είμαστε έτοιμοι να γίνουμε αξιόπιστοι γιατί όταν γίνονται ασκήσεις ε, ε, είναι στην ουσία μια ένδειξη που δείχνει ότι δεν πρέπει να τολμήσεις να κάνεις το δεύτερο αυτό δημοψήφισμα. Δεν θέλω ξαφνικά να έχω πρασινοφορεμένους στα μέσα της Ευρώπης. Ε, πρέπει λοιπόν να δράσουμε και γιατί έχουμε προληπτικά μέτρα και δρόμους, ε, ε, να δούμε δηλαδή κατά πόσο είμαστε σε ετοιμότητα για να σταματήσουμε κάτι τέτοιο με το στρατό. Ευχαριστούμε τον Μίχαλ Κάλερ. Κύριε Σκουζή, έχουμε τώρα λίγα λεπτά χρόνια για να απαντήσετε στις ερωτήσεις, ε, γιατί μετά θα έρθουν οι συνάδελφοι από τις δύο άλλες επιτροπές. Ευχαριστώ, Έντουερτ, και για την ερώτηση και για τα λουλούδια. Όπως έχει επιβεβαιώσει η Ιμφοστάτη υπάρχουν διαφορές ε, στη Ρεπούμπλικα σέρπστικα και την Ομοσπονδία που έχουν επιβεβαιωθεί από την Ιμφοστάτη. Κύριε Πίτσολα, κάποιες φορές επειδή δεν έχουμε χρόνο ε, πρέπει να, απλοποιούμε. Εγώ θα ήθελα λιγότερο Dayton και περισσότερο Βρυξέλλες. Όμως οι Βρυξέλλες πρέπει να είναι ισχυρές. Δεν πρέπει να υπάρξει κενό εξουσία στη Βοσνία Ριζεγοβίνη. Πρέπει να είμαστε εκεί μαζικά. Η προτεραιότητα τώρα. Ποιες προτεραιότητες μετά από τόσα χρόνια στην Βοσνία Ριζεγοβίνη το κράτος δικαίου είναι το σημαντικό. Γιατί έχουμε στην Ρουμανία ε, τόσα άτομα στη φυλακή, γιατί είναι πολύ ισχυρό ο εισαγγελέα. Το ίδιο πρέπει να γίνει και στη Βοσνία Ριζεχοβίνη. Δεν είναι μόνο τα οικονομικά ζητήματα, είναι και το κράτος δικαίου που παίζει ρόλο. Κύριε Ράντο, οι συνταγματικέ συναποφάσεις είναι τώρα δεσμευτικές και ε, οι 29 υπάρχουν τώρα, οι 20 δεν έχουν εφαρμοστεί ακόμα. Έτσι λοιπόν πρέπει να δούμε την σχέση, αλλά όπως και να έχει, κάθε απόφαση του συνταγματικού δικαστηρίου που δεν εφαρμόζεται είναι κρίμα. Γιατί το συνταγματικό ε, δικαστήριο δεν αποφασίζει και το θέμα αν θα το εφαρμόσεις ε, είναι στη διακριτική σου ευκαιρία, ευχέρεια. Είναι υποχρέωση για όλους. κάποιες ερωτήσεις ε, για τον εκλογικό νόμο, ειδικά για την περίπτωση Γιουζίτς ε, πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος. Να πω ότι πρέπει να αλλάξει και σε πολιτικό επίπεδο. Υπάρχουν ανάγκες που πρέπει να αντιμετωπιστούν, αλλά πρέπει να αλλάξει με συνένεση. Δεν έχουμε, ας πούμε, ε, κάλπες γυάλινες ε, στη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Ε, ας πούμε στην Εστονία έχουν ηλεκτρονική ψηφοφορία, θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Υπάρχουν πολλές βελτιώσεις που μπορούν να γίνουν για να μπορεί ο κόσμος να ψηφίζει. Αλλά σίγουρα το θέμα είναι κυρίως πολιτικό και υποστηρίζω σίγουρα την πρόθεση. Αν υπάρχουν τρεις λαοί στην Βοσνία Ερζεγοβίνη, ε, ε, όταν είμαστε αδέρφια πρέπει να φροντίζουμε το μικρότερο αδελφό. Όλοι έχουν δικαιώματα, αλλά κάποιοι άλλοι έχουν λίγο περισσότερα ε, ε, στο χαρτί για να αισθάνονται καλύτερα. Δεν υπάρχει δίλημα γι' αυτό από τη δική μου πλευρά. Κύριε Φρόιντ, ναι, πιο ισχυρός ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για άλλη μια φορά το κράτος δικαίου είναι το κλειδί. Πρέπει να γίνουν πολλά, αλλά η Βοσνία Ριζεγοβίνη είναι στο σωστό δρόμο. Ε, πρέπει να δείξουμε ότι το θέμα είναι κατεπήγον. Δεν μπορεί να είναι απλώς μια γραφειοκρατική διαδικασία όπως ήταν και στις άλλες χώρες. Λειτουργήσε στη Βαλτική, αλλά στα Βαλκάνια δεν λειτουργεί αυτή η διαδικασία. Πρέπει να βάλουμε και κάποιο πολιτικό επίγον στην διαδικασία. Και, ναι, το αν θα δεχτούμε τη Βοσνία Ερζεγοβίνη με τα λάθη της, ναι. Έτσι είναι, ως υποψήφια όμως, όχι ως κράτος μέλος. Γιατί ε, όταν είσαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχεις υποχρεώσεις, πρέπει να κάνεις πιο πολλά και πιο γρήγορα. Και μεταξύ της υποψηφιότητας ε, και της ε, ημέρας της ένταξης υπάρχει αυτή η διαδικασία λουκάνικο που τη λέμε. Όπως καταλαβαίνετε αυτή η μετάβαση, η μεταβατική περίοδος είναι το πιο σημαντικό. Ε, κύριε Βάγκλερ, λυπάμαι. Στην ε, Βοσνία Ερσεγοβίνη τα σύμβολα ε, χρησιμοποιούνται υπέρ των δέων. Είτε είναι για, στη μνήμη κάποιας, κάποιου γεγονότος, αλλά γενικά στο Βερολίνο, για παράδειγμα, η Γερμανία, έχει κάτι αντίστοιχο. Κάθε πέντε μέτρα στο Βερολίνο βλέπεις ένα μνημείο. Όμως η Γερμανία είναι μια ισχυρή χώρα παρόλα αυτά και προοδευτική. Ε, τώρα, ε, ε, μπορούμε να αναπτύξουμε τη χώρα και οι νέοι να είναι ε, ευγνώμονες. Οι πολιτικοί πρέπει να δουλέψουν περισσότερο για το μέλλον. Φυσικά η ακαδημαϊκή και ο πολιτισμός, αλλά πρέπει να μείνουν οι νέοι εκεί. Ε, όπως είπε ο υπουργό, το 70% των νέων θέλουν να δουλέψουν για κρατικές εταιρείες όπως η Telecom, αλλά επίσης θέλουν να βγουν και στο εξωτερικό το 70% των νέων. Τώρα, όταν είσαι χριστιανός, ε, είναι καλό να είσαι γενναιόδωρος. Ε, οπότε Φέτος, οπωσδήποτε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το έτος. Το χρόνο έχουμε τις εκλογές όπως είπε και ο κύριος Τσενάρκ, ε, πρέπει να υπάρχει συνδυασμένος κύκλος εκλογών, γιατί αλλιώς έχουμε συνεχώς προεκλογική περίοδο, συνεχώς νεοσχηματιστήσεις κυβερνήσεις. Είχαμε τρεις εκλογές σε τέσσερα χρόνια και είναι σημαντικό να συντονίζουμε την εθνική και τις τοπικές εκλογές, ε, γιατί αλλιώς δεν υπάρχει χρόνος να δουλέψεις εν ειρήνη. Ε, τώρα, ποιο είναι το χειρότερο σενάριο. Δεν θέλω να το σκεφτώ. Αν υπάρξει τάση από τη Ρεπούμπλικα Σέρψκα να αποσχιστεί, φυσικά θα έχουμε πρόβλημα ε, δεν θέλω όμως καν να το σκεφτώ. Εγώ απλώς σας ζητώ κάθε φορά που έχετε τη δυνατότητα να ψηφίζετε υπέρ της επέκτασης της εντολής της U4 που είναι μια ιστορία επιτυχημένη, έχει κάνει πολύ καλή δουλειά, δεν είναι τόσο δαπανηρή, δεν συμφωνούν όλες οι χώρες, αλλά εγώ την υποστηρίζω στεναρά, έχει συμβολική η, ε, η παρουσία της. Από τις 600.000 πήγαμε στα 600 άτομα. Όμως είναι μια ε, συνεκτική δύναμη. Δίνει ασφάλεια στον κόσμο ότι δεν θα γίνει κάποια νέα σύραξη. Τώρα για τα ποσοστά δεν έχω κάποια νούμερα καινούρια, αλλά είναι γύρω στο 60 80% υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστούμε κύριε Ίσκο που ήρθατε στην Επιτροπή μας. Ευχαριστούμε που απαντήσατε σε όλα μας τα ερωτήματα. Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο Σαράγεβο. Και τώρα κλείνουμε την συνεδρίαση. Η επόμενη συνάντηση είναι στις 2 Μαΐου το πρωί και το απόγευμα και 3 Μαΐου το πρωί στις 9 μέχρι τις μισή. Τώρα, παρακαλώ. Γεια σας.